Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και θα αφιαρίσω λίγο ε, μέχρι να έρθουν κάποια κάποιοι ακόμη. Θέλω λοιπόν να σας καλωσορίσω όλες και όλους θερμά στην ε, σημερινή μας ε, συνεδρίαση. Καταρχάς, για να εγκρίνουμε το σχέδιο μερισιάς διάταξης, θέλω να ρωτήσω αν συμφωνείτε όλοι με το σχέδιο μερισιάς διάταξης. Δεν βλέπω να υπάρχει κάποια αντίρρηση. Επομένως, θεωρώ ότι εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Ερχόμαστε στο δεύτερο σημείο της διάταξη, διάταξης, έγκριση των πρακτικών των συνεδριάσεων. 22 και 23 Μαρτίου έχετε το σχέδιο λέει Μάρτιος βέβαια, αλλά κανονικά έπρεπε να είναι Μάης. Α, όχι, Μάη, Μάρτης. Ω, πέρασε τόσο καιρό. Άρα, 22-23 Μαρτίου έχετε το σχέδιο των πρακτικών στο φάκελό σας. Υπάρχουν παρατηρήσεις, υπάρχουν αντιρρήσεις. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Προτείνω λοιπόν, όσοι ήθιστε, να θεωρήσουμε ότι είναι εγκεκριμένα τα πρακτικά εφόσον δεν θα έχουμε ενημερωθεί για κάποια αντίρρηση μέχρι το τέλος της σημερινής συνεδρίασης. Ερχόμαστε τώρα στο σημείο της, ε, το 3 που είναι η ανακοινώσει της Προέδρου. Σήμερα έχουμε διερμηνία στις εξής γλώσσες. Γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, τσεχικά, εστονικά, πολωνικά, ουγγρικά, σλοβενικά, βουλγαρικά, ρουμανικά. Πρέπει να σας ενημερώσω επίσης ότι η συνεδρίαση αυτή μεταδίδεται και στο διαδίκτυο και σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις ε, των συντονιστών της 21ης Ιουνίου, τις λάβατε με email στις 23 Ιουνίου και θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται εφόσον δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας της 28ης Ιουνίου η οποία και έλξε, άρα θεωρούμε ότι έχουν εγκριθεί. Επίσης, ε, έχουμε τη συνάδελφα η εξελέγει στη ε, Βουλή και δεν μπορεί να είναι εδώ από την ομάδα ECR συντονίστρια. Θέλω λοιπόν να, να καλωσορίσω τον, ε, μάλλον συγχαρώ τον συνάδελφο Τζαμπάσκι που θα αντικαταστήσει συνάδελφο από το ECR και ελπίζω να συνεργαστούμε καλά. Ο κύριος Στογεύσκη επίσης μου ζήτησε να του δώσω σύντομα το λόγο για να μας ενημερώσει, για, αν κατάλαβα καλά, για μια εκδήλωση σήμερα το μεσημέρι με την Ομοσπονδία, με την αντιπροσωπεία της Λευκοσίας. Παρακαλώ, πείτε μας. Ναι, ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Γνωρίζω ότι Υπάρχουν συνάδελφοι που ενδιαφέρονται για τις εξελίξεις στη Λευκοσορία. Στο PHS στις 2 σήμερα έχουμε την επίσκεψη ε, μια ομάδα εργασίας για τα θέματα που απτονται της Λευκορωσίας. Ε, ουσιαστικά πρόκειται για τη διαδικασία της Μπολόνια ε, και την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας. Στην συνάντηση αυτή θέλουμε να μιλήσουμε και για τα πλεονεκτήματα, αλλά και για τις δυσκολίες που προκύπτουν στη Λευκορωσία από την εφαρμογή της διαδικασίας αυτής. Δύο η ώρα λοιπόν στο PHS. Σας ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος, μας ενημερώσατε για την εκδήλωση αυτή. Εντάξει, πέρασε λίγο η ώρα, ήρθαν και άλλοι συνάδελφοι, οπότε νομίζω τώρα μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 4, που είναι η ώρα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και συγκεκριμένα έχουμε την ψήφιση της ε, εκθέσεως ιδέας πρωτοβουλία σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας του Κοινοβουλίου και Συμβουλίου με μερμή 13 Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με την καταπολέμηση σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. Συγγήτριά μας ήταν η Ζαμπίνε Φερχάιν. Θες να πεις κάτι σύντομα, κυρία Φερχάιν, ναι, πολύ σύντομα. Θέλω να πω ότι συνεργαστήκαμε εξαιρετικά με τους γιώδες συζητητές και τους υπόλοιπους συναδέλφους. Ήταν και άκρως υποδομητικές οι τροπολογίες. Θέλω να ευχαριστήσω επίσης και τη Φαμπιά για την πάρα πολύ καλή συνεργασία που είχαμε. Και νομίζω ότι πλέον έχουμε μια πολύ καλή γνωμοδότηση για την Επιτροπή Λίμπε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και όλους τους συναδέλφους. Θα ευχαριστήσουμε και την Φαμπία που πηγαίνει στο Ταλίν και γι' αυτό δεν μπορεί να είναι εδώ σήμερα. Θα τις μεταφέρουμε τι ευχαριστίες σου πάντως και μπορούμε τώρα να περάσουμε τι στην ψηφοφορία και αρχίζουμε με τη συμβαστική ένα υπέρ. Κατά απόχέ, εγκρίνεται. Τροπολογία 9 υπέρ. Κατά απόχέ. εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική ε, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται.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 Τροπολογία 34 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 35 υπέρ, κατά, θα ελέγξουμε, ναι. Άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται 11 υπέρ, 11 κατά, ισοψηφία. 36 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές από 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελέγχουμε και αυτήν. Την 38 λοιπόν. Ελέγχουμε. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 13 ψήφοι υπέρ, 9 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 39 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 40 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 47 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στην τροπολογία 56. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 64 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 66 υπέρ κατά αποχές θα ήθελα να ελέγξουμε την 66 παρακαλώ έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 11 προς 10. Εγκρίνεται. Τροπολογία 67 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 68. Δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Ορίστε. Α, ναι, πρέπει να πω ότι υπάρχει και προφορική τροπολογία εδώ. Το ξέχασα. Στο δεύτερο τμήμα υπάρχει λοιπόν προφορική τροπολογία. Δεν ξέρω, το έχετε στον κατάλογό σας. Μήπως πρέπει κάποιος να μας το αιτιολογήσει. Η Σίλβια μήπως βέβαια γνωρίζουν περί τίνος πρόκειται. Kann ich mal bitte Μήπως κανείς μπορεί να μας αναγνώσει την προφορική τροπολογία. Είναι από την ομάδα Σοσιαλιστών και Δημοκρατών που αφορεί και αυτή τροπολογία. Σίλβια. Αυτή η τροπολογία προβλέπει την ακύρωση της τελευταίας στο δεύτερο τμήμα των λόγων των λέξεων Internet Service Providers Συγγνώμη, αλλά δεν το βρίσκα. Δηλαδή η διαγραφή στο τέλο αυτή τη παραγράφου του δεύτερου τμήματο, εκτός από αυτές τις λέξεις που θέλουμε να διαγραφούν. Ωραία, είναι σαφές. Υπάρχει κάποιο που να αντίθεση με αυτήν την προφορική τροπολογία. Από ό,τι φαίνεται όχι, επομένω μπορούμε να ψηφίσουμε. Αλλά παρακαλώ να τις ε, καταθέτεται εγκαίρω για να μπορούμε να τι έχουμε και στους καταλόγους της προφορικής τροπολογία. Λοιπόν, δεύτερο τμήμα τη 68 με την προφορική τροπολογία ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 69 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχέ. Εγκρίνεται 70 υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 75 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 83 υπέρ, κατά, αποχές, θα ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 83. Πέρας. 12 κατά, 10 υπέρ, απορρίπτεται. Τροπολογία 84 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 85 υπέρ, με προφορική τροπολογία. Κύριε Φερχάν, ουσιαστικά είναι γλωσσικής φύσεως. Urges the member states to introduce in the legislation volunteering for activities and jobs Δηλαδή, end for activities and jobs και το και έλειπε. Για δραστηριότητες και θέσει εργασία. Ωραία, δεν υπάρχει κάποιος που αντίθετος. Ψηφίζουμε λοιπόν μαζί με την προφορική των 85 υπέρ, κατά, αποχές. Η ομάδα των Σοσιαλιστών Κρατών τι ήταν, υπέρ ή κατά. Ich mach das Παναλαμβάνουμε την ψηφοφορία. Ποιοι είναι υπέρ, κατά, Ωραία. Εγκρίθηκε. 86 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στην τροπολογία 94 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 95 υπέρ κατά αποχές θα ήθελα να ελέγξουμε. 95 άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. 13 υπέρ 9 κατά εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 99 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 108 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πηγαίνουμε στην τροπολογία 110 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 111 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 112 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται Ερχόμαστε τώρα, τώρα στην τελική ψηφοφορία που θα είναι με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Geschlossen. Πέρασε ψηφοφορία. 22 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά. Με μεγάλη πλειοψηφία έγινε δεκτή η νομοδότηση και θέλω να συγχαρώ τη συντάκτα της νομοδότησης, την κυρία Φερχάη. Παρακαλώ όσοι θέλουν να αποχωρήσουν, παρακαλώ ησύχω ε, και τάχιστα να το πράξουν. Δεν ξέρω πού βρίσκεται ο εμπειρογνώμονας, ίσως έχει μείνει στην κίνηση, έχει κολλήσει. Μάρτιν, μη φύγεις. Η πρότασή μου θα ήταν, λοιπόν, να προτάξουμε το σημείο 6 που είναι ο Γενικός Προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί αν βλέπω σωστά είναι παρόντες όλοι και οι εισηγητές οπότε νομίζω ότι μπορούμε να συζητήσουμε πρώτα το 6 για να μην χρειαστεί να διακόψουμε τη συνεδρίαση μας εφόσον συμφωνείτε βέβαια. Ωραία, επομένως περνάμε στο σημείο 6 της Μέσης Διάταξης Γενικός Προπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Οικονομικό έτος 2018 όλα τα τμήματα Και εδώ έχουμε την εξέταση του σχεδίου γνωμοδότηση που συνέταξε ο συνάδελφό μα Μόρτεν, συγγνώμη, Λεκεγκάρτ, στον οποίο θα δώσω και ευθύ αμέσω το λόγο. Μόρτεν, Έχει το λόγο, So, Ευχαριστώ, αγαπητοί συνάδελφοι. Λίγα πράγματα θα ήθελα να πω για τη θέση της Επιτροπής μας για το Γενικό Προϋπολογισμό της Ένωσης για το Οικονομικό έτος 2018. Είχαμε κάνει μια γενική συζήτηση την περασμένη εβδομάδα. Την Δευτέρα ήταν η προθεσμία για την κατάθεση των τροπολογιών. Θα ήθελα να σας δώσω κάποιες λεπτομέρειες για τη διαδικασία. Η Γραμματεία της Επιτροπής μας έχει λάβει 47 τροπολογίες συνολικά και έχουμε προτάσεις και για τα πιλωτικά προγράμματα και για τις προπαρασκευαστικές δράσεις, ε, για τις βασικές δημοσιονομικές γραμμές. Δεν έχω μπει σε λεπτομέρειες, δεν είχα την δυνατότητα να τις διαβάσω όλες λεπτομερώς, όμως... Ε, Ελπίζω ότι μέχρι αύριο θα έχετε ε, όλες τις τροπολογίες, ε, η γραμματεία δηλαδή θα σας τις ε, διανύμει, μπορεί να τις περιμένετε δηλαδή αύριο. Έχουμε μια συνάντηση σκιωδών την επόμενη Τετάρτη στο Στρασβούργο, κατά την οποία βάσει των καλών συζητήσεών μας ως τώρα Πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε καλές συμβιβαστικές τροπολογίες. Θα προτείνω κάποιες βασικές γραμμές για το Erasmus ε, Plus ε, για, κατά τη συνεδρίασή μας ε, των σκιωδών την Τετάρτη όσον αφορά τα πιλωτικά προγράμματα και τις προπαρασκευαστικές δράσεις. Ο στόχος μου είναι να ακολουθήσω τη μακροχρόνια πρακτική της Επιτροπής μας να υποστηρίξουμε τις, ε, τις τροπολογίες ε, που ε, έχουν λάβει ένα α ή ένα β τουλάχιστον, αν θυμάμαι καλά, ότι συνήθως υποστηρίζουμε τις α, αλλά θα δούμε ότι όταν θα μπούμε στις διαπραγματεύσεις, όταν θα έχουμε δηλαδή τον κατάλογο μπροστά μας, θα το δούμε πιο συγκεκριμένα. Για την ώρα δεν έχω λάβει απολύτως τίποτε, θα το δούμε όταν θα λάβουμε το πλήρη κατάλογο το χρονοδιάγραμμα είναι πάρα πολύ ε, στενό 6 ε, του μηνός ε, είναι η, ε, μάλλον έξι ώρα τη Δευτέρα είναι η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών και την Τετάρτη θα συναντηθούν οι σκιώδεις όπως είπα προηγουμένως. Θέλουμε πάντως να περάσουμε κάποια βασικά μηνύματα στο πλαίσιο της Επιτροπής μας. Θα θέλα να υπάρξουν, να προτείνω εγώ κάποιους συμβιβασμούς την επόμενη Τετάρτη. Νομίζω ότι είχαμε ήδη πολύ καλές συζητήσεις την περασμένη εβδομάδα για τις γραμμές προϋπολογισμού. Ελπίζω να έχετε χρόνο να εξοικειωθείτε με τις τροπολογίες. Θα σας δώσω μόνο γενικές πληροφορίες ε, για τη λογική μου, ε, τη λογική της προσέγγισής μου από τότε που συναντηθήκαμε. Πρώτο σημείο, μετά τις ε, συζητήσεις με τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την περασμένη φορά, άκουσα και τις, ε, δικής του, τις δικές τους συστάσεις. Ζητούμε επιπλέον 50 ε, ε, εκατομμύρια για το Erasmus Plus στο πλαίσιο του EMFF από το 2016 στο 2020 και θέλουμε να έχει ολοκληρωθεί η εκταμείευση του ποσού μέχρι το 2018. Θέλουμε κατανομή αναλογική 44 εκατομμύρια στην εκπαίδευση και στην κατάρτιση και 6 εκατομμύρια στα επιμέρους προγράμματα για την νεολαία. Γνωρίζω ότι κάποιοι άλλοι έχουν προτείνει μία κατά τη διαφορετική κατανομή. Εγώ ευχαρίστω να δω και άλλη αναλογία κατανομής του κόστους. Δεύτερο σημείο, έχουμε ακόμη κάποιες ανησυχίες για τον προϋπολογισμό στο σώμα, ως προς το σώμα αλληλεγγύης, γιατί αντλεί μεγάλο ποσοστό χρηματοδότησης από το Erasmus Plus και θέλουμε ακόμη κάποιες απαντήσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Παρόλο που μας εγγυήθηκαν ότι θα αφορά μόνο το πρόγραμμα EVS, το πρόγραμμα εθελοντικής ε, ε, υπηρεσίας. Ε, δεν βγαίνουν τα νούμερα ακόμη και στη γνωμοδότηση εγώ θα επιμείνω ότι κανένα άλλο ποσό εκτός από αυτό του EVS δεν θα φύγει από το Erasmus Plus για να πάει στο σώμα αλληλεγγύης. Όσον αφορά την υποχρηματοδότηση των επιμέρους προγραμμάτων για τη δημιουργική Ευρώπη και την Ευρώπη για την νεολαία, προτείνω επιπλέον 2 εκατομμύρια ευρώ για τις διευκολύνσεις αυτές και συμφωνώ με, τις, με τα 14 εκατομμύρια αύξηση που προτείνει ο για οι δημοκράτες για τη δημιουργική Ευρώπη. Τέταρτον, ε, για τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς του 2018, συμφωνώ με το να επιμείνουμε σε μια ξεχωριστή γραμμή προπολογισμού, ε, ώστε τα 7 ε, εκατομμύρια να είναι εμφανή στον προϋπολογισμό. Και επίσης, σημείο 5, όσον αφορά τις δράσεις για τα μέσα. Ε, εγώ ήρθα σε επαφή με συναδέλφους ε, ως προς το θέμα αυτό. Ε, ελπίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ε, δώσει τα 2 εκατομμύρια ε, για το 2018. Βέβαια αυτό είναι μια μείωση από τα 6 εκατομμύρια του 2016. Είναι μικρότερο το ποσό. Επομένως στην γνωμοδότηση θα ζητήσουμε ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασφαλίσει μια βιώσιμη μακροχρόνια λύση ώστε το πρόγραμμα αυτό να είναι ένα μόνιμο πρόγραμμα το οποίο θα μπορούσε ε, να χρησιμοποιεί σωστά τα κονδύλια του, να δαπανώνται δηλαδή σε σωστές δράσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, με χαρά αναμένω τις ε, επερχόμενες συζητήσεις που θα λάβουν χώρα την Τετάρτη. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε Μόρτεν. Τώρα θα ήθελα να δώσω το λόγο στους σκιώδεις εισηγητές. Παρακαλώ να δηλώσετε ποιοι θέλετε να μιλήσετε. Ο κύριος ε, Στρογεύσκη είναι ο πρώτος. Δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Με πολύ συγκεκριμένο τρόπο υποδείξατε τις προτεραιότητες και ε, χαίρομαι γιατί η συνεργασία με τον εισηγητή είναι εξαιρετικά σημαντική και είναι ήδη πολύ θετική. Ωστόσο διαβλέπω μία δυσκολία καθώς έχουμε δύο κείμενα παράλληλα και ένα πρόγραμμα Πρόκειται για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι το 2020 και έχουμε τώρα τον προπολογισμό για το 2018 όπου βλέπουμε πράγματα ανησυχητικά. Το τρίτο στοιχείο είναι το, στοιχείο, το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Δεν ξέρω πού θα βρούμε ε, τα 50 εκατομμύρια για το Erasmus Plus, τα οποία έχουν ανακοινωθεί παλιότερα, ενώ ταυτόχρονα προτείνεται να χρηματοδοτηθεί το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. με ε, τα χρήματα αυτά του Erasmus ε, Plus. Και αυτό δεν μπορούμε να το δεχτούμε, γιατί πρώτον δεν έχουμε μέσα, μιλάμε για τους πόρους και στο επόμενο έγγραφο ακριβώς ε, βλέπουμε αυτό, αυτό το ποσά και ότι αυτό το ποσό θα φύγει από το Erasmus Plus. Εγώ πιστεύω πως ο στόχος ε, του Erasmus Plus δεν είναι το ίδιο με το ίδιο μάλλον με αυτούς τους Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία, ε, όπου υπάρχουν επικαλύψεις, αλλά δεν είναι 100% τα ίδια. Οι ίδιοι στόχοι. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να δεχτούμε την αφαίρεση πόρων από το Erasmus Plus. Τώρα, ε, όσον αφορά το ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν εδώ πολύ ανησυχητικά στοιχεία γιατί μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις στις πληρωμές. Εάν παραμείνουμε στις, ε, στα προγνωστικά για τις πληρωμές και τα εξετάσουμε, βλέπουμε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν τα ίδια προβλήματα που είχαμε πριν δύο χρόνια. Όσον αφορά δηλαδή τις πληροχωρώσεις και τις πληρωμές. Ε, εγώ νόμιζα πως αυτό το πρόβλημα το είχαμε λύσει πριν κάποια χρόνια, ενώ τώρα βλέπω πως επανέρχεται. Euronet, 2 εκατομμύρια. Στην ουσία πρόκειται για απόλυτη εξάλληψη και εκμηδένιση αυτού του προγράμματος. Κυρίες και κύριοι, στην Ολομέλεια είπαμε ότι οι ευρωπαϊκοί θεσμοί οφείλουν να καταπολεμήσουν την προπαγάνδα και την παραπληροφόρηση. Οφείλουμε να αγωνιστούμε κατά αυτού του είδους τα, των ε, γεγονότων. Και το Euronet Sin είναι ένα εκπαιδευτικό μέσο, ένα εργαλείο μέσω του οποίου ενημερώνουμε για το τι εργασίες κάνουν οι θεσμοί. Και αν υπάρξει εδώ περικοπή, είχαμε 6 εκατομμύρια και τώρα 2. Οπότε η κατάσταση είναι εξαιρετικά σχετική. Παλιότερα η κατάσταση ήταν διαφορετική, ενώ ταυτόχρονα θέλουμε να στηρίξουμε τις δράσεις στο πλαίσιο της ε, πληροφόρησης για τον ε, πολιτισμό. Τώρα γνωρίζουμε όλο ένα και περισσότερα πράγματα. Θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε 100% πρέπει να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να αυξήσουμε τις γνώσεις. Γιατί οι γνώσεις είναι οι πιο σημαντικές για την παιδεία, για τους νέους και για τα παιδιά. Εκτός μικροφώνου. Ε, <clears throat> Grazie Presidente, ringrazio innanzitutto il relatore per σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ τον εισηγητή πρώτα απ' όλα για την έκθεση που μας έχει υποβάλει και θα κάνω ή κάποιες κύριες παρατηρήσεις και στη συνέχεια βεβαίως τα υπόλοιπα θα τα δείτε με τις τροπολογίες που θα τα, τις δείτε την επόμενη εβδομάδα. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω στα όσα μόλις ε, αναφέρθηκαν ε, και τονίστηκαν την ιδέα δηλαδή που έχουμε και εμείς υπογραμμίσει με την ευκαιρία της προηγούμενης συνεδρίασης για τα 100 εκατομμύρια που προβλέπονταν για το εράσμος Plus στην αναθεώρηση του PDP. Αυτό ήταν ε, το νούμερο. Και άρα το αίτημα είναι να ανακτήσουμε αυτό που προβλεπόταν από το PDP. Ε, ε, διαπιστώνουμε ότι θα υπάρξει ε, επιστολή και πιθανότατα διορθωτικός προϋπολογισμός που τουλάχιστον θα καλύπτει 50 εκατομμύρια που είχαν μείνει, αλλά τα 50 ήδη είχαν χορηγηθεί για το 2017. Θεωρώ ότι τα επιπλέον 50 δις, ε, εκατομμύρια συγγνώμη, και εδώ το λέω για τον εισηγητή, πιθανότητα θα πρέπει να δρομολογηθούν για φέτος για να ευθυγραμμιστούμε με τις απαιτήσει, αλλά και για να αντισταθμίσουμε τον αντίκτυπο του σώματος αλληλεγγύης στο Erasmus Plus. Θεωρώ πως δεν είναι καθόλου σκόπιμο να επικαλεστούμε την ανάγκη επένδυσης στους νέους και μετά να μετρα... μειώνουμε τον προϋπολογισμό ε, που τους έχουμε αφιερώσει. Και, και απλά σε συμβολικό επίπεδο πιστεύω πως το μήνυμα αυτό είναι τελείως λανθασμένο. Γι' αυτό και θεωρώ ότι θα ήταν σκόπιμο να ανανεώσουμε στο κείμενο του γνωμοδότησης μια υπενθύμηση της σημασίας της επένδυσης στην πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Χωρίς όμως να ξεχνάμε ότι πρέπει να στηρίξουμε την εσωτερική ζήτηση ώστε να δημιουργήσουμε ε, ανάπτυξη και απασχόληση. Ε, να πω επίσης ότι προβληματίζομαι όσον αφορά την νέα ε, το νέο προγραμματισμό για την ε, προετοιμασία για την Ευρώπη στον τομέα νέων του Erasmus Plus. Εκεί προβλέπεται ο περιορισμός των κονδυλίων για το σώμα αλληλεγγύης και επίσης να δημιουργηθεί μια προπαρασκευαστική δράση που δεν προβλέπεται που θα χρειαζόταν και νομική βάση και δικούς της πόρους. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί μας δίνεται η εντύπωση σε αυτή τη φάση ότι το Erasmus Plus θεωρείται ένα είδος omnibus όπου χωρίς καμία σαφήνεια πλέον ε, λειτουργεί ο τομέας των νέων ως ένα ε, σκουμπαράς ε, από όπου παίρνει ο καθένας ό,τι χρειάζεται. Εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να επανέλθουμε στα όσα ορίστηκαν στο ΠΔΠ. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Η Χέλγα Τρούπελ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ευχαριστώ και τον Μόρτεν για την παρουσίασή του. Εγώ συμφωνώ με, τους, με τις φιλοδοξίες σας για την ε, αύξηση της χρηματοδότησης ε, της δημιουργικής Ευρώπης ε, και της Ευρώπης για τους πολίτες, για να υπάρχει μεγαλύτερη προώθηση και ορατότητα, επίσης και για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Τώρα, όσον αφορά το Σώμα Αλληλεγγύης, υπήρξε το αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην χρησιμοποιηθούν χρήματα από το Erasmus Μετά υπήρξε η πρόταση ε, βάσει της οποίας ε, υπόθηκε ότι ναι, ε, ακούμε την πρότασή σας και παίρνουμε χρήματα μόνο από την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, από το EVS, που είναι τμήμα του Erasmus+, για να ε, είναι, να, να, να προσθεθούν στη νέα ε, προσέγγιση και το νέο προϋπολογισμό για ε, το σώμα αλληλεγγύης. Όμως τα 20 εκατομμύρια τελικά τα παίρνουμε από το Erasmus Plus για το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης που δεν συνδέεται άμεσα με την Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία και νομίζω ότι πρέπει να ξέρουμε αν αυτό είναι ε, όντως ισχύει και αν ισχύει τότε ε, πρέπει να πούμε ότι ναι μεν ε, πήραμε τα χρήματα από την Εθελοντική Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, αλλά δεν υπήρξε επιπρόσθετο ποσό. Ναι, είναι πολύ καλή ιδέα το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, αλλά δεν θα έπρεπε να ε, ζημιώνει αυτό κάποια χρήματα τα οποία είχαν πρικοδοτηθεί για το Erasmus Plus, που δεν συνδέεται άμεσα με το Σώμα Αλληλεγγύης για τα επιπλέον... 50 εκατομμύρια. Ναι, πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό το ποσό και εμεί ω πράσινοι υποβάλαμε πρόταση πώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον προπολογισμό τη επόμενη χρονιά και πώ να κατανεμηθούν. Όμω για το σώμα αλληλεγγύη πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Νομίζω ότι ε, και η πλειοψηφία είναι υπέρ τη προσπάθεια αυτή να δοθούν ευκαιρίε στου νέου ανθρώπου σε ολόκληρη την Ευρώπη, όχι όμω ζημιώνοντα τον προπολογισμό του Erasmus Plus ε, όλα τα χρήματα δηλαδή που είχαν αφιερωθεί ειδικότερα ε, στο Erasmus Plus για όλα αυτά τα χρόνια. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Δεν νομίζω ότι... Α, όχι, υπάρχει ακόμα κάποιος που θέλει το λόγο. Η Σίλβια Παρακαλώ. Ευχαριστώ τον εισηγητή και τους κοιόδες, γιατί πιστεύω ότι έχουν πραγματικά συμβάλει επί της ε, σαφούς βάσης που έδωσε ο συνάδελφος για να μιλήσουμε για αυτή μας την ε, θέση. Και θέλω λοιπόν να επαναλάβω τα εξής. Το πρώτο είναι ότι για τον πολιτισμό το αίτημα που είχαμε κάνει και με τις τροπολογίες μας ήταν ακριβώς ότι λόγω της υποτίμησης του προβλήματος media και του Κουλτούρα να έχουμε 14 ε, παραπάνω για το Μέντια και 11 παραπάνω για το Κουλτούρα. Γιατί διαφορετικά θα ήταν ε, ανεπαρκή η πρόταση. Έπειτα, ε, συμμερίζομαι την πρόταση να επαναλάβουμε ότι θα πρέπει να αποκατασταθούν τα 50 εκατομμύρια γιατί αυτό προβλέπει το, η πρόταση της Κομισιόν για το 2018 και ότι θα πρέπει να αποσαφινιστεί, όπως έλεγε η Χέλγα Τρούπελ, από το ε, ΣΒΕΤ που τώρα παίρνουμε σε μόνο σε αυτή τη μεταβατική περίοδο τα χρήματα. Αυτό ήταν και η πρόταση της Κομισιόν, θα πρέπει αυτό να το καταστήσουμε σε θέση στην έκθεσή μου. Και θα ήθελα επίσης να έχω κάποιες παραπάνω πληροφορίες για το θέμα καταλάβω καλύτερα αν ε, ε, πρόκειται τώρα για προπαρασκευαστική δράση που περνάει στο δεύτερο ή τρίτο χρόνο της, για... Ε, δεν θα μπορεί να μπει σε συγκεκριμένη γραμμή του προϋπολογισμού ή αν θα έρθει αυτό μόλις ολοκληρωθεί το... η τριετία. Αυτό θέλω να ρωτήσω από τον Λόκιμπεργκ. Ακόμα μια παρατήρηση και τελειώνω για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Θα πρέπει να είναι σαφές ότι τα περίφημα 4 εκατομμύρια, 1 για το 17 και 3 για το 18 αφορούν ακριβώς την συγκεκριμένη αύξηση. Τα υπόλοιπα όμως δεν θα πρέπει να είναι στους πόρους για το ε, ευρωπαϊκό έτος. Μας μένουν μόνο 3 για φέτος από αυτά τα εκατομμύρια. Σας ευχαριστώ. Νομίζω ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό συμφωνούμε όλοι εδώ στην Επιτροπή μας ότι πρέπει να στείλουμε ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα με την γνωμοδότησή μας ε, και την έκθεση μας προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε σχέση με το Erasmus Plus, ότι δεν θέλουμε να ε, χαθούν κονδύλια από το Erasmus ε, για το σώμα αλληλεγγύης, ενώ ήδη ε, και για την εθελοντική υπηρεσία ε, που προβλέπονταν κάποια χρήματα μπορεί και αυτά να αφαιρεθούν. Δεν θέλουμε λοιπόν ε, να ζημιωθεί αυτό το κονδύλι του προϋπολογισμού. Και σε ό,τι αφορά την επαγγελματική κατάρτιση, Εκεί επίσης έχουμε κάποια δείγματα ότι θα φύγουν κάποια κονδύλια και θα πάνε στο σώμα αλληλεγγύης και νομίζω ότι πρέπει η δική μας Επιτροπή να στείλει ένα πολύ ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν είμαστε διατεθειμένοι να δεχθούμε κάτι τέτοιο και από ό,τι βλέπω στην Επιτροπή μας υπάρχει μεγάλη συνένεση ως προς αυτό. Να δώσω πάντως το λόγο για μια ακόμη φορά στον ε, Μόρτεν Λόκεγκορτ για την προθεσμία. 3 Ιουλίου στι 4 το μεσημέρι, μα το είπε βέβαια ήδη, να παραλάβω αυτή την προθεσμία για την κατάσταση τροπολογιών. Την Τετάρτη την προσεχή στο Στρασβούργο υπάρχει συνάντηση των σκιωδών εισηγητών για να συζητηθούν οι τροπολογίε που θα έχουν κατατεθεί, όπως συμφωνήσαμε, στα αγγλικά, λόγω τη πάρα πολύ σύντομη προθεσμία. Δεν θα ήταν λογικό. Ε, διαφορετικά δεν θα προλάβαιναν οι σκιώδεις. Ε, Α, η Κομισιόν, επειδή το προτάξαμε το θέμα αυτό, ε, δεν είναι και αυτή εγκαίρος εδώ, ε, ε, κόλλησαν και αυτοί, τέλος πάντων. Βέβαια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκάθαρα δηλώσε ότι εφόσον υπάρχουν ερωτήματα, μπορούν είτε τηλεφωνικός είτε γραπτός να τα απαντήσουν. Ε, ο Μόρτεν έχει ξανά το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ και όπως πολύ σωστά είπατε, ε, διαισθάνομαι μεγάλη ομόνια μεταξύ των συναδέλφων της Επιτροπής μας για το θέμα αυτό, οπότε δεν θα σχολιάσω πολύ περισσότερο. Από ό,τι καταλαβαίνω, ε, μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν υπάρχουν ε, ιδιαίτερες ανησυχίες σε σχέση με τα 15 εκατομμύρια. Αν κατάλαβα καλά, αυτά τα χρήματα όντως ε, θα ε, δοθούν. Το θέμα είναι πώς ακριβώς θα κατανεμηθούν. Και βεβαίως θα το συζητήσουμε αυτό όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης και εγώ τις ίδιες ανησυχίες με εσάς έχω συνάδελφοι και κατά τη γνώμη μου αυτό θα είναι ο μεγάλος αγώνας ε, φέτος, κατά πόσο δηλαδή πώς θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το γεγονός ότι δεν μεταφερθούν χρήματα από το Erasmus Plus εδώ πιστεύω ότι θα παραμείνουμε ενωμένοι. Ε, τουλάχιστον αυτό κατάλαβα από τα σχόλια που άκουσα. Όσον αφορά τώρα το ερώτημα της κυρίας Κώστα, εγώ είχα κάποια προβλήματα με την ε, μετάφραση, μήπως θα μπορούσαμε διμερώς ε, να το συζητήσουμε μετά, γιατί πρέπει να καταλάβω ακριβώς τι, μου, τι με ρωτήσατε. Δεν κατάλαβα ακριβώς τι ακριβώς θέλετε να πείτε. Θα το σημειώσουμε βεβαίως και θα το συζητήσουμε μετά. Νομίζω ότι είμαστε ενωμένοι, συμφωνούμε και με πολύ χαρά αναμένω τις συζητήσεις μας την επόμενη Τετάρτη. ευχαριστώ πολύ Μόρτεν. Κάθε επιτυχία σε σένα και στους σκιώδεις εισηγητές. Το έχει δείξει και το παρελθόν όμως ε, ότι ό,τι έχει να κάνει με τον προϋπολογισμό ιδίως ε, ε, είναι θέματα τα οποία μας βρίσκουν σύμφωνους. Υπάρχει, θα έλεγα, ομοφωνία μεταξύ των μελών της Επιτροπής, οπότε δεν φαντάζομαι να προκύψουν προβλήματα. Τουλάχιστον στη δική μας Επιτροπή. Δεν ξέρω, έχω κάποιες αμφιβολίες για το τι θα γίνει αν χρειαστεί να δώσουμε μάχη με την Κομισιόν και το Συμβούλιο. Να περάσουμε τώρα ένα βήμα πίσω, γυρίζοντας τη μέση διάταξη, στο σημείο 5 Έχουμε την παρουσία της μελέτης που είχε ζητήσει η Επιτροπή μας από το Τμήμα Πολιτικής Ο τίτλος της μελέτης ήταν «Διδασκαλία κοινών αξιών στην Ευρώπη». Τον Ιανουάριο του 2016 συγκεκριμένα είχαμε ζητήσει από το θεματικό αυτό τμήμα να καταρτήσει την εν λόγω μελέτη, η οποία πλέον είναι έτοιμη και μπορεί σήμερα να μας ε, παρουσιαστεί. Και θέλω λοιπόν να καλωσορίσω θερμά τον κύριο Βιλ Φόγκελερς από το Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών της Ουτρέχτης. Θα τον παρακαλέσω σύντομα, δηλαδή για 10 λεπτά, ε, να μας παρουσιάσει τα πορίσματα της μελέτης αυτή. Κύριε Φόγκελερς, καλώς ορίσατε. Good morning everybody. I will speak in English. Καλημέρα σας. Ε, Ολλανδικά είναι η μητρική μου γλώσσα, αλλά θα σας τα πω στα αγγλικά. Καλημέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε την, μου δίνετε τη δυνατότητα να σας παρουσιάσω τη μελέτη μας. Today I will present Σήμερα θα σας παρουσιάσω το πρόγραμμα διδασκαλίας των κοινών αξιών, πώς δηλαδή τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβάνουν τις αξίες της δημοκρατίας και της ανεκτικότητας στις ε, εφαρμοζόμενες εκπαιδευτικές πολιτικές. Εγώ είμαι καθηγητής ε, ε, εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Ανθρωπιστικών Σπουδών του Σουτρέχτης στις κάτω χώρες, στην διακήρυξη των Παρισίων ε, οι Υπουργοί Εκπαίδευσης ζήτησαν περισσότερη εστίαση ε, της εκπαίδευση στη διδασκαλία κοινών αξιών όπως η δημοκρατία και η ανεκτικότητα. Αυτές οι δύο αξίες θεωρούνται βασικές ε, αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημά μας, ε, στο οποίο βασίστηκε η έρευνα, ήταν το εξής. Ε, ποια είναι η πολιτική εκπαίδευση και η πρακτική ε, διδασκαλίας κοινών αξιών δημοκρατίας και ανεκτικότητας στις 28 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα χρησιμοποιώ από εδώ και στο εξής το ακρονίμιο TCV. Ε, δύο μελέτες κάναμε. Πρώτον, μία μελέτη πολιτικής εκπαιδευτικής σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα 28 και ε, συζητήσαμε με ακαδημαϊκούς εμπειρογνώμονες του τομέα και επίσης έγινε και μία μελέτη του προγράμματος σε 12 χώρες. Ε, ουσιαστικά είδαμε δηλαδή την πρακτική που ακολουθείτε και κάναμε και κάποιες συνεντεύξεις. Οι μελέτες αυτές οι μεμονωμένες έχουν συμπεριληφθεί στην μελέτη μας. Θα ήθελα να πω μερικά πράγματα για το ενοιολογικό μας πλαίσιο. Το ενοιολογικό πλαίσιο της μελέτης μας βασίστηκε σε δύο έννοιες. Το πρώτο ήταν αυτό της δημοκρατίας. Έγινε μία διάκριση, μία αναφορά σε τρία στοιχεία. Πολιτική συμμετοχή, ε, δημοκρατικές, ε, δημοκρατική πολιτική και δημοκρατική ε, κοινωνία. Μία ελεύθερη, χωρίς αποκλεισμούς, κοινωνία. Επίσης, το στοιχείο της ανεκτικότητας, ε, δύο είδη ανεκτικότητας, η ίδια προσωπική ανεκτικότητα, η ανεκτικότητα προς άλλα κοινωνικά και άλλες κοινωνικές και πολιτιστικές ομάδες και στο πλαίσιο της κοινωνίας. Προσπαθήσαμε να δούμε τις επιρροές της εκπαιδευτικής πολιτικής ε, στα σχολεία, για παράδειγμα. Ε, υπήρχαν κάποια ζητήματα που αφορούσαν για παράδειγμα ε, την εκπαίδευση για την ε, ιδιότητα του πολίτη, κάποιες, κάποια άλλα μαθήματα που αφορούσαν την ιστορία, τη γεωγραφία και επίσης τη μεθοδολογία, την κουλτούρα και την, το πόσο μεγάλη είναι η διαφορετικότητα. Κάναμε τη διάκριση μεταξύ των στόχων, των μέτρων και της αυτονομίας σε επίπεδο πολιτικής και σε επίπεδο ε, πλαισίου είδαμε ε, τη συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων και της ευρύτερη κοινότητας. Να περάσω τώρα στα αποτελέσματα. Ποια είναι τα αποτελέσματα των ε, μελετών μας. Υπάρχει μια αυξημένη προσοχή στη διδασκαλία των αξιών της δημοκρατίας και της ανεκτικότητας, κάτι που είναι προφανές στις εκπαιδευτικές πολιτικές όλων των κρατών μέλων της Ένωσης. Η διδασκαλία των αξιών αυτών είναι σημαντικό τμήμα της εκπαίδευσης στο ίμιση των κρατών μελών, ε, όμως ε, σε σχέση με άλλους τομείς του επιστητού, η προσοχή σε αυτές τις αξίες δεν είναι επαρκής. Ε, τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσουν έναν έντονο διάλογο ως προς το τι ακριβώς είναι αυτές οι κοινέ αξίες και ποιος είναι ο ρόλος της εκπαίδευσης και επίσης τα κράτη-μέλη πρέπει να ενισχύσουν την ανάπτυξη οράματος ε, ιδεών ε, καινοτόμων πολιτικών, πρακτικών όπως επίσης και ανταλλαγή καλών παραδειγμάτων και εμπειριών. Όσον αφορά την εφαρμογή της πολιτικής, πώς ε, εφαρμόζεται η πολιτική για τη διδασκαλία κοινών αξιών. Τα κράτη-μέλη της Ένωσης ε, διαφοροποιούνται στον τρόπο με τον οποίο ε, καθοδηγούν την διδασκαλία των κοινών αξιών. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ του σχολικού προγράμματος και των συγκεκριμένων μέτρων, δηλαδή κατευθυντηρίων γραμμών κλπ. Υπάρχει επίσης και ένα χάσμα μεταξύ ε, των ε, στόχων και των ε, μέτρων. Τα αποτέλεσμα λοιπόν είναι ότι πολλές φορές τα σχολεία δεν δίνουν επαρκή προσοχή στη διδασκαλία των κοινών αξιών. Μερικά σχολεία χρησιμοποιούν την αυτονομία τους, αλλά όχι. Οι συστάσεις μα λοιπόν σε σχέση με την εφαρμογή διδασκαλίας των κοινών αξιών είναι το ότι η καθοδήγηση ε, πρέπει να είναι πιο ε, καλή και να ε, εστιάζεται κυρίως γενικούς στόχους και τις κατευθυντήριες γραμμές και θα πρέπει επίσης τα σχολεία να ε, ενθαρρύνονται να δώσουν μεγαλύτερη προσοχή ε, στις αρχές της δημοκρατίας και της ανεκτικότητας. Τι γίνεται τώρα στα σχολεία, ποια είναι η πρακτική. Το ίμιση των κρατών μελών έχουν μάθημα, ε, κάποιο είδους μάθημα ηθικής ή εκπαίδευση για την ιδιότητα του πολίτη. Σε μερικά σχολεία αυτό συμπεριλαμβάνεται στην ιστορία, αλλά δεν στοχεύεται ειδικά η εκπαίδευση στους τομείς της δημοκρατίας και της ανεκτικότητας ε, ή υπάρχουν κάποιες άλλες παράπλευρες δραστηριότητε που δεν είναι τμήμα του σχολικού προγράμματος. Ε, άλλα ε, σχολεία έχουν πιο ιδεολογική προσέγγιση. Υπά, όσο υπάρχει κάποια συμμετοχή των ε, σπουδαστών, αλλά δεν υπάρχει δημοκρατική κουλτούρα στα περισσότερα σχολεία. Υπάρχουν κάποιοι δεσμοί με την κοινότητα και τι μη κυβερνητικέ οργανώσει, αλλά αυτοί οι δεσμοί δεν είναι πάρα πολύ ισχυροί συνήθω και προτείνουμε τα κράτη-μέλη να ενθαρρύνουν ολοκληρωμένη χρήση όλων αυτών των ε, στοιχείων για, ώστε η διδασκαλία των κοινών αξιών να βελτιωθεί όντως. Η σχέση μεταξύ του σχολείου και του εξωτερικού κόσμου ε, μπορεί να γίνει ε, ισχυρότερη με την ενίσχυση του δεσμού με την κοινότητα και τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Όσον αφορά τώρα τις έννοιες, ε, μια εκπαιδευτική πρακτική ε, πρέπει εστιάζεται στην πράξη στη συμμετοχή λιγότερο στην δημοκρασία, στη δημοκρατία ε, και στην ανάπτυξη ε, συνένεσης η ανεκτικότητα επικεντρώνεται ε, στα διάφορα επίπεδα πολιτιστικών ομάδων, αλλά λιγότερο στην κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς. Εμείς προτείνουμε τα εξή ε, στα σχολεία ε, και στα κράτη-μέλη. Να δοθεί προσοχή σε όλα τα στοιχεία της δημοκρατίας και της ανεκτικότητας. Είναι σημαντική η γνώση, αλλά η ανάπτυξη μιας δημοκρατικής και ανεκτικής νοοτροπίας είναι επίσης πάρα πολύ σημαντική. Η έννοια της ανεκτικότητας, η έννοια της ε, ε, ε, συμμετοχής με σεβασμό είναι επίσης πολύ σημαντική στο πλαίσιο της ανεκτικότητας. Και για να ολοκληρώσω, τα πορίσματά μας τα τελικά είναι ότι υπάρχει ένα χάσμα μεταξύ των στόχων, των προθέσεων και των μέτρων στο επίπεδο της πολιτικής. Υπάρχει επίσης ένα χάσμα μεταξύ πολιτικής και πρακτικής και υπάρχουν και διαφορές μεταξύ των χωρών. Οι συστάσεις μας ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη είναι οι εξή. Βελτιώσεις σε όλα τα στοιχεία της διδασκαλίας των κοινών αξιών, δημοκρατίας και ανεκτικότητας. Υπάρχουν ενδιαφέροντα παραδείγματα και υπάρχουν πολλές ε, δυνατότητες καινοτόμων πρακτικών ε, πρέπει να ενισχυθεί στα σχολεία η ανταλλαγή ε, εμπειριών και πρακτικών και μεταξύ των σχολείων ώστε να ενισχυθεί η διδασκαλία κοινών αξιών. Το μέλος του κόσμου μας ε, χρειάζεται μια ισχυρή εστίαση ε, στις αξίες, σε κοινέ αξίες όπως η δημοκρατία και η ανεκτικότητα. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Φόγκελες για την παρουσίαση της μελέτης σας που νομίζω ότι ότι μας δίνει πολύ χρήσιμα στοιχεία για το μελλοντικό μας έργο. Μου έχουν ζητήσει ήδη το λόγο κάποιοι συνάδελφοι, τον οποίο πρώτος ο κύριος Σβέρ. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο κύριε Πρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω κύριε Φάγκελερς για την παρουσίαση της μελέτης και για την έρευνα Χαίρομαι πολύ που έχουμε αυτή τη μελέτη, γιατί το έλεγα και το ξανά έλεγα τα προηγούμενα χρόνια. Δεν έχουμε έρευνα ε, στον τομέα αυτό. Και πιστεύω πραγματικά πως ε, η κοινή πολιτιστική μας κληρονομιά είναι και ο ισχυρότερος δεσμός που ενώνει τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πολιτισμός ε, συνδέει, μας φέρνει πιο κοντά, πολύ περισσότερο από ότι ο χάλιβας ή τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Η Ευρώπη έχει κοινή πολιτιστική κληρονομιά. Περί πρόκειται όμως. Αυτή η κοινή πολιτιστική κληρονομιά βασίζεται στη χριστιανική πίστη, στην ε, ρωμακαθολική παράδοση, στην ελληνική φιλοσοφία, στο μοντερνισμό. Επίσης έχουμε κοινέ αξίες στην κοινή μας ιστορία. Κυρίως τη δημοκρατία και την ανεκτικότητα. Είναι αξίες, αλλά είναι και πολιτικές αρχές. Και βέβαια υπάρχει και η αλληλεγγύη, ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, η ειρήνη, η ευημερία, η ισότητα μεταξύ των φίλων. Αυτές είναι βασικές αξίες από τον οποίο δράση η Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να τις ε, προασπίζεται. Και ακόμη και αν έρχονται άλλοι ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν ε, έχουν την ίδια πολιτιστική παράδοση και δεν σέβονται τη δική μας ε, πρέπει να προσπίσουμε την δική μας παράδοση. Μιλήσατε για τα σχολεία και είπατε ότι έχουν ένα βασικό ρόλο, ένα ρόλο κλειδί. Δεν είναι μόνο τα σχολεία, πρέπει και τα μέσα επικοινωνία και γενικότερα την πολιτική σφαίρα να την ε, ενσωματώσουμε, όπως και τις οικογένειες τους γονείς, τους νέους. Οι νέοι ουσιαστικά ανατρέφονται από τους γονείς τους. Ε, από αυτούς παίρνουν τις βασικές αρχές και αξίες, αλλά και τα σχολεία σίγουρα είναι πολύ σημαντικά. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να, ασκήσουν κάποια επιρροή στα σχολεία. Μέχρι στιγμής υπήρχε άποψη ότι τα σχολεία ε, θα πρέπει να είναι ουδέτερα ως προς την ε, μεταλαμπάδευση αξιών. Δηλαδή δεν πρέπει να μεταφέρουν τα σχολεία κάποιες αξίες, αλλά ε, θεωρώ αντιθέτως ότι τα σχολεία μπορούν και πρέπει να έχουν έναν ενεργητικό ρόλο για να διαμορφώνουν την κοινή γνώμη στις κοινωνίες μας και πιστεύω ότι μπορούν να αναδείξουν και να βελτιώσουν τη δημοκρατική κουλτούρα που είναι και προϋπόθεση για τη σωστή λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών. Και πάλι ευχαριστώ για τη μελέτη σας. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ πολύ. Το λόγο τώρα έχει η κυρία Κώστα. Εξαιρετικά σημαντική αυτή η έρευνα βέβαια, γιατί ξεκινά από τη βούληση να δούμε ε, τι συμβαίνει στις διάφορες χώρες, ε, στις παιδαγωγικές τους μεθόδους σε σχέση με τα προγράμματα τα εκπαιδευτικά και στους τρόπους με, τον τους οποίους ε, ε, εισάγουν το θέμα των ε, αξιών στις, ε, στην ύλη. Να πω τα θετικά στοιχεία, να δούμε μετά και τα πιο αρνητικά για να έχουμε ένα διάλογο. Ενδιαφέρον είναι ότι κάνατε μια ανάλυση που ελέγχει από το, ότι από τη ε, δεκαετία του 90 και μέχρι σήμερα έχει δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στα κράτη-μέλη και στα προγράμματα τα κατευθυντήρια και τις γραμμές της κατευθυντήριας για την ε, αγωγή του πολίτη. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που μας λέτε ε, αρχικά ενδιαφέρον για να καταλάβουμε πώς ε, η ευρωπαϊκή διάσταση θα πρέπει να συνοδεύει την εθνική. Ο ορίζοντας είναι πολύ εθνικός. Ενώ εμείς θέλουμε να αναζητήσουμε τις αξίες, της κοινέ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάποια κράτη-μέλη έχουν εντοπίσει χωριστά αυτό το θέμα και άλλα όχι. Και έπειτα το θέμα των προτάσεων που δίνεται για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να προωθήσουμε ανοίγοντας τα σχολεία και στις εξωτερικές σχέσεις, ας πούμε στο Ιταλικό σύστημα, προβλέπονται εξωσχολικές διαδικασίες που συνδέονται με την δράση του πολίτη, τις αξίες ε, του, της αλληλικής κτλ. Μπορούμε να κάνουμε και εκπαιδευτικές πιστώσεις, αν ένα παιδί ας πούμε, ασχολείται με τον εθελοντισμό, με την ε, ενεργή δηλαδή αλληλεγγύη. Εσείς ξεκινήσατε να ορίσετε κοινέ αξίες μετά τη δήλωση ε, των Υπουργών μετά από την τρομοκρατική, τις τρομοκρατικές επιθέσεις που, επίσης, που βασίζονται στη δημοκρατία και στην ανοχή. Εγώ πιστεύω πως πρέπει να ανοίξουμε λίγο τον ορίζοντα. Δεν πιστεύω πως η ανοχή λύνει όλα τα προβλήματα ελληνικής και ειρηνική συμβίωση. Θα έπρεπε να έχουμε δηλαδή ένα πιο ευρύ φάσμα θεμελιωδών αξιών, δηλαδή ελευθερία, αξιοπρέπεια του ατόμου, ε, διεθνή συνεργασία πέρα από την δημοκρατία και την ανοχή. Αυτή λοιπόν η έρευνα εστιάζεται σε αυτό, είναι δική σας επιλογή γιατί χρειάστηκε να ξεκινήσετε από κάπου. Εγώ είχα την εντύπωση ότι θα μπορούσε να είναι μια ευκαιρία, επειδή ακριβώς σήμερα αμφισβητώνται ε, τα εκπαιδευτικά συστήματα που ίσως να εδράζονται στη δημοκρατία και την ανοχή, αλλά δεν μιλάνε για ε, δυνατότητες ε, ενό σχολείου για όλους. Εσείς το τονίζετε και με χαροποίησε που ορισμένε χώρες όπως και η δική μου δίνουν προσοχή στο ένταξη, για παράδειγμα, των ατόμων με ειδικέ ανάγκες ή των μεταναστών. Αυτό το θέμα της διαπολιτισμικότητας επίσης δεν έχει τονιστεί καθόλου. Ίσως λοιπόν να είναι μια βάση για να μπούμε σε βάθος και να διευρύνουμε το φάσμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία ε, ίσως δύσκολα σημεία, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμα για τη συζήτηση. Έβλεπα ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα για ένα χωριό στην Ουγγαρία και την πολιτική του Όρμπαν, που έλεγε ξεκάθαρα ότι ακολουθεί την αρχή της εθνικής ομοιογένειας, κάτι που για μένα δεν ευθυγραμμίζεται με αυτό που εμείς εννοούμε όταν μιλάμε για δημοκρατία και ανεκτικότητα, διότι η ανεκτικότητα σημαίνει πάντοτε ότι έχει να κάνει με διαφορετικέ μειονότητε, αλλά είσαι ανοιχτό απέναντί του. Έχει μεν τι αξίε σου, αλλά προσπαθεί να βρει ένα κοινό παρονομαστή κατανόηση για να αντιμετωπίσει αντιπαραθέσει όχι ότι αφήνει εκτό ε, τμήματα κοινωνία που μπορεί να προέρχονται από άλλο πολιτιστικό υπόβαθρο, να έχουν άλλη θρησκεία και ούτω καθεξής. Δεύτερο, ένα άρθρο στην Τσάι Zeitung από μια αναλυτρία, την κυρία Κρίστεβα, διάβασα, το οποίο ήταν πολύ ξεκάθαρο και μίλα για το πρόβλημα των ευρωπαϊκών αξιών στη Γαλλία. Και μιλούσε για νέους Αλγερινούς, Αλγερινού υποβάθρου νεαρούς Γάλλους και έλεγε ότι υπάρχουν μεγάλα προβλήματα στη Γαλλία, διότι η κοινωνία στη Γαλλία δεν αντιμετώπισε με το σωστό τρόπο τον πόλεμο της Αλγερίας ε, και τα πιο κρατικά ε, θέματα, την απεικιοκρατική ιστορία. Η Γαλλία πρέπει να το αυτό το πρόβλημα, να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της Αλγερίας και της απεικιοκρατίας, γιατί αυτοί οι νέοι που είναι μεν Γάλλοι υπήκοοι δεν νιώθουν Γάλλοι. Νιώθουν οι Αλγερινείς αυτής καταγωγής, Αλγερινής καταγωγής αυτοί νέοι ε, Γάλλοι ότι είναι εκτός της κοινωνίας. Γι' αυτό και πολλές φορές ε, κάποιοι καταφεύγουν μέχρι και στην τρομοκρατία. Όλο το ζήτημα λοιπόν της ανεκτικότητας είναι πολύ σημαντικό. Ιδίως όταν υπάρχουν τμήματα της κοινωνίας που δεν έχουν ε, ταυτιστεί με τη χώρα στην οποία ζουν, δεν νιώθουν ότι ανήκουν σε αυτήν. Σίγουρα ε, υπάρχουν και σφάλματα και από την πλευρά των μεταναστών. Το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει προσπάθεια ε, συνεννόησης. Επίσης, είχαμε και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πριν κάνα μήνα για... Είχαμε και ένα ραβίνο εδώ που μίλησε για τον αντισημιτισμό. Είπε ότι δεν είναι το βασικό πρόβλημα για του Εβραίου. Φυσικά και είναι πρόβλημα γιατί έχουν υποφέρει. Αλλά ουσιαστικά είναι πρόβλημα για τι κοινωνίε εν γέννη. πρέπει να είναι ε, ανοιχτές και να μπορούν να αντιμετωπίσουν τη διαφορετικότητα. Αλλιώς δεν είναι αξιόπιστες και δεν μπορούν να ε, συμπεριφερθούν σωστά. Και όταν μιλάμε εδώ τώρα για τη διδασκαλία κοινών αξιών, νομίζω ότι και στα σχολεία αλλά και σε άλλους φορείς ε, και στην πολιτική συζήτηση είναι πολύ σημαντικό να βρούμε τρόπο ώστε να συμμετέχουν σε αυτό το διάλογο άνθρωποι από διάφορα, διαφορετικά υπόβαθρα. Δεν σημαίνει ότι είναι σωστοί αυτοί που ακούμε συνήθως ε, που έχουν τη δυνατότητα να μιλούν. Απλά πρέπει να υπάρχει αυτό το ανοιχτό πνεύμα. Αυτή είναι η βάση για μια ανοιχτή κοινωνία. Πρέπει να ακούμε τι απολυτικέ. να υπάρχουν αντιπαραθέσει, μπορεί να υπάρχουν συγκρούσει, αλλά και αυτό γόνιμο είναι. Η ανταλλαγή καλών πρακτικών είναι κάτι θετικό. Απλά σε κάποιο βαθμό θα έλεγα ότι χρειάζεται να αλλάξουμε νοοτροπία. Πώ να το πω. Να το δούμε αλλιώ. Και αυτό είναι το ερώτημα. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις συγκρούσεις που μπορεί να προκύπτουν ή πρέπει να τις ε, βάλουμε κατά από το χαλί. Δεν είναι ρεαλιστικό κάτι τέτοιο. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να κάνουμε να συμμετέχει ο κόσμος πιο επικοδομητικά και είναι ένα ερώτημα για όλους. Σε ευχαριστώ πολύ Χέλγκα. Δύο ακόμη έχουν στήσει το λόγο. Τρεις. Και μετά θα κλείσω τον κατάλογο των ομιλητών. Κυρία Σόντροβα είναι επόμενη. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση τη μελέτη αυτή και η έρευνα ήταν πάρα πολύ σημαντική. Κοίταξα τα στοιχεία για την Τσεχία, γιατί είμαι από την Τσεχία. Και πρέπει να σας πω ότι η μελέτη αυτή πραγματικά είναι πολύ σημαντική γιατί έχετε πραγματικά περιγράψει με πολύ εύγλωτο τρόπο το τι γίνεται στην Τσεχία, πώς γίνεται αυτή η διδασκαλία των κοινών αξιών στην Τσεχία. Και αυτό που μου έκανε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν η πολύ σωστή παρατήρηση που κάνατε, ότι δηλαδή θα πρέπει στις τάξεις να προσφέρεται ένα ασφαλές περιβάλλον για να συζητούνται αυτές οι κοινέ αξίες. Και γι' αυτό πραγματικά ε, χρειάζεται δουλειά ακόμη ε, και ότι πρέπει να συζητούμε επίκαιρα ζητήματα στα σχολεία. Και επίσης η συστηματική επιμόρφωση των καθηγητών, των εκπαιδευτικών. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η ε, εκπαίδευση των εκπαιδευτών, η προετοιμασία τους, η επιμόρφωσή τους ε, έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε σχέση με αυτά τα θέματα που συζητούμε. Έχω μια ερώτηση. Στην παρουσίασή σας επαναλαμβάνετε την ε, απέτηση ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών που έχουν αποδειχθεί επιτυχημένες και αυτό να γίνεται από τα σχολεία, από τα καθηγητές, από τα κράτη-μέλη. Κατά την άποψή μου, αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ε, στοιχείο ε, που θα προωθήσει την ανταλλαγή κοινών αξιών. Γιατί εκεί μπορούμε να δούμε τις βασικότερες και πιο επιτυχημένες μεθόδους των κρατών μελών και να υπάρξει μίμηση αυτών των μεθόδων από άλλους. Ε, Μίλησε και η Χέλγα Τρουπέλ για τις ε, κοινέ αξίες ε, και το ερώτημα είναι ακριβώς αυτό. Πώς θα πετύχουμε να διαδάξουμε, να μεταλαμπαδεύσουμε αυτές τις κοινέ αξίες, στις κοινωνίες μας ε, στα κράτη-μέλη της Ένωσης και ξεχωριστά σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να αναλύσουμε και να εξετάσουμε το πώς εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε από το ευρωπαϊκό επίπεδο τα κράτη-μέλη να προωθούν τις κοινέ αξίες στα σχολεία, στη νέα γενιά. Και εδώ θα ήθελα να σας κάνω το εξής ερώτημα. Ποια εργαλεία κατά την απόψή σας είναι τα πιο σημαντικά για αυτό το σκοπό. Ευχαριστώ. Η πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Μάλινοφ. Thank Σας ευχαριστώ για τη μελέτη και για την παρουσίαση. Όπως ε, καταλαβαίνετε είναι πολύ εύκολο να μιλάμε και να επικρίνουμε για αυτό το θέμα. Γιατί είναι τόσο γενικό και όριστο. Εγώ θέλω να πω δύο λόγια. Εκτός ίσως του πλαισίου αυτής της συζήτησης, αλλά είναι κάτι που με ενοχλεί ανέκαθεν όταν έχουμε ε, τέτοιε μελέτες για τις κοινέ αξίες και βλέπω πάλι το ίδιο πράγμα. Η δημοκρατία είναι ένα πολιτικό καθεστώς, είναι μια διαδικασία. Το παράδοξο όταν μιλάμε για την δημοκρατία ως αξία είναι ότι είναι λάθος. Η δημοκρατία είναι μια διαδικασία, είναι, διαδικασία, ε, είναι, ε, ε, ένα σύστημα, ένα πολιτικό καθεστώς. Ανάλογα με τις αξίες μιας δημοκρατικής κοινωνίας, το δημοκρατικό καθεστώς μπορεί να λειτουργήσει με διαφορετικούς τρόπους. Μπορεί να λειτουργήσει και οδηγεί σε ανελεύθερες δημοκρατίες, μπορεί να οδηγήσει σε απολυταρχισμό και επί τη βάση των αξιών μπορεί να οδηγήσει σε κάτι που εννοούμε όταν λέμε δημοκρατία. Για μένα λοιπόν το να διδάξουμε αξίε σημαίνει να διδάξουμε αυτές τις αξίες που ε, κάνουν τη δημοκρατία να λειτουργεί. Όχι απλά να λέμε ότι η δημοκρατία είναι καλή. Γιατί μετά κάποιοι από αυτού του νέου θα ανακαλύψουν ότι η δημοκρατία μπορεί να συνδυαστεί και με τον ρατσισμό ε, και μπορεί να βρεθούν σε μειονεκτική θέση και τότε να είναι αντιδημοκρατική και να ριζοσπαστικοποιηθούν. Κατά τη γνώμη μου λοιπόν οι αξίες θα πρέπει να οριστούν πιο συγκεκριμένα. Αξίες όπως η ελευθερία, η αλληλεγγύη, η αξιοπρέπεια, η ισότητα των φύλων και μετά να δούμε πώς αυτά λειτουργούν στις διάφορες χώρες που ε, ισχυρίζονται ότι είναι δημοκρατικές και να δούμε τις διαφορές. Είμαι βέβαιος ότι η ισότητα των φύλων δεν είναι πρόβλημα στις περισσότερες χώρες. αλλά στις ευρωπαϊκές χώρες εννοώ. Άλλου είδους όμως ανισότητες εμφανίζονται και βλέπετε ότι η ισότητα σημαίνει πολύ διαφορετικά πράγματα για τον καθένα. Η αξία αυτής της προσέγγισης είναι ότι βλέπεις πραγματικά πού έγκυται οι δυσκολίες, οι αδυναμίες σε κάθε χώρα. Εγώ μπορώ να πω ότι σε αρκετές χώρες πρώην κομμουνιστικές υπάρχει πολύ συγκεκριμένη απαξίωση αυτών των ε, ε, ε, αξιών. Και γι' αυτό και η δημοκρατία δεν είναι σταθερή. Και επίσης κάτι που εγώ είδα στην πράξη που λειτουργούν είναι οι διαφορετικές διδακτικές μέθοδοι. Αυτό είναι της αξίας. Καθώς επίσης η συμμετοχή των νέων σε διάφορες μορφές δημοκρατικής διαδικασίας, ενώ είναι ακόμα στο σχολείο ή στο πανεπιστήμιο. Ακόμα και μέθοδοι υπάρχουν για τις ακόμα χαμηλότερες, μικρότερες ηλικίε. Είναι πολύ διαφορετικό και αντιμετωπίζονται διάφορα είδη ελλημάτων αξιών για την δημοκρατία. Μάλιστα θα επέμενα για ένα πολύ, πολύ συγκεκριμένο σχόλιο, δηλαδή διδασκαλία μεθόδων αξιών και όχι διδασκαλία αξιών. τελευταίος ομιλητής. Δεν θέλω, να... Δεν θέλω να ε, μεταφέρω σε άλλη κατεύθυνση το διάλογο, ωστόσο θα ήθελα να αντιδράσω, γιατί όταν λέτε ότι ο Βίκτορ Όρμπαν μιλάει για εθνοτική ομοιογένεια, σαφώς αναφέρεται στη μετανάστευση. Γιατί, φέρτε μου ένα άρθρο εφημερίδας παρακαλώ, γιατί αν ο Βίκτορ Όρμπαν μιλά για εθνοτική ομοιογένεια, μιλά για την μετανάστευση. Είναι μια σπουδαία αξία κατά, κατά να υπάρχει μια ισχυρή Ευρώπη των εθνών. Θέλουμε αυτό να διατηρηθεί. Βεβαίω οι μετανάστες πρέπει να ε, να τους μετανάστες και τους πρόσφυγες πρέπει να τους υποδεχτούμε, αλλά το 90% ε, των, προσφύγων δεν είναι πρόσφυγες, είναι οικονομικοί μετανάστες. Μπορούμε να μιλήσουμε για την μετανάστευση, μπορούμε να μιλήσουμε για το πώς θα τη σταματήσουμε, αλλά το πρόβλημα το μεταναστευτικό, κατά τη γνώμη μου, θα πρέπει να σταματήσει στη Λιβύη. Εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να πάω σε άλλη κατεύθυνση και σέβομαι το θέμα, αλλά έπρεπε οπωσδήποτε να αντιδράσω σε αυτή την παρατήρηση. Ωραία. Να παρακαλέσω τώρα αν ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να μιλήσει σε σχέση με τη μελέτη αυτή. Ε, θέλετε. Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Σίλβια Κάλμα λέγομαι και είμαι από τη Γενική Διεύθυνση εκπαίδευση και Πολιτισμού. Ε, συντονίζω το φάκελο για την ε, διακήρυξη των Παρισίων. Θα ήθελα εκ μέρους τη Επιτροπής να επικροτήσω την ε, μελέτη την οποία ανέδεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι πάρα πολύ επίκαιρη η δημοσίευσή, η της γιατί βρισκόμαστε εν μέσω προβληματισμού για ένα συγκεκριμένο εργαλείο ε, για την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και την ε, προώθηση των κοινών αξιών μέσω της, επίθυμη, της επίσημης ε, μάθησης. Έχουμε επίσης και μία διαβούλευση σχετικά με το ρόλο της εκπαίδευσης για την προώθηση των κοινών αξιών. Θα ήθελα να σας ενθαρρύνω να συμμετέχετε κι εσείς και να το διαδώσετε και στους εμπλεκόμενους φορείς και στις περιφέρειές σας. Μπορεί να θέλουν να συμμετέχουν. Έχουμε λάβει πάνω από 200 απαντήσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης αυτής. Η διαβούλευση κάνει ερωτήσεις ε, δύσκολες, ε, ε, ποιες είναι οι πιο αποτελεσματικές πρακτικές για την ενθάρρυνση των κοινών αξιών και της κοινωνικής ένταξης και πώς μπορούν τα κράτη-μέλη να το επιτύχουν αυτό με τον καλύτερο τρόπο. Η σύσταση του Συμβουλίου, την οποία επεξεργαζόμαστε, προγραμματίζεται για το τέλος του 2020 και ο στόχος της σύστασης θα είναι ακριβώς ε, η εδραίωση ε, το, της γνώσης που έχουμε για το θέμα αυτό και η παροχή υποστήριξη στα κράτη-μέλη σε σχέση με το πώς θα καταφέρουν τους στόχους. Έχετε αναφέρει ήδη κάποια σημαντικά στοιχεία στο πλαίσιο της μελέτης σας. Είναι γεγονός ε, ότι η, η διδασκαλία των κοινών αξιών, η διδασκαλία δεν μου αρέσει βέβαια πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να διδάξει κανείς αξίες, γιατί οι αξίες ε, πρέπει να ε, τις μαθαίνει κανείς μέσω εμπειρίας. Υπάρχουν πολλές, πολλά στοιχεία όπως το σχολικό πρόγραμμα, η προετοιμασία των δασκάλων που μπορεί να συνεισφέρουν σε αυτό. Αναφέρατε επίσης ε, σε ένα ασφαλές δημοκρατικό περιβάλλον σχολικό, ε, η ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών. Υπάρχουν πάρα πολλοί τομείς που ε, υπησέρχονται και προσπαθούμε να αποκρισταλώσουμε αυτή τη δουλειά. Υπάρχει και μία ομάδα εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο της ατζέντα για το 2020 που εργάζεται ειδικά για την προώθηση των αξιών και ε, της ε, μη διακριτικής μεταχείρισης μέσω της εκπαίδευσης. Ε, συμμετέχουν εμπλεκόμενοι φορείς όπως μη κυβερνητικέ οργανώσεις, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών, διεθνείς οργανώσεις, στο πλαίσιο πολιτικής για να προωθηθούν οι κοινέ αξίε και η κοινωνική ένταξη και υπάρχει μάλιστα και ένα οδηγό στο διαδίκτυο ε, προ αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ για την μελέτη σα. Βλέπω ότι τα συμπεράσματά σα ε, συμβαδίζουν με τα δικά μα και εμεί συλλέγουμε κάποια στοιχεία. Υπάρχει το νέο δίκτυο EDC ε, ε, για την ε, εκμάθηση της ε, ιδιότητας του πολίτη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχε μία έκθεση ήδη από το 2012, αλλά θα υπάρξει άλλη μία, η οποία θα δημοσιευθεί το φθινόπωρο, γιατί κάνει μία ανάλυση σε όλες τις χώρες Τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα να αναφερθώ και στην έκθεση του Συμβουλίου της Ευρώπης που δημοσιεύθηκε πριν από μερικές μέρες για την κατάσταση τη εκπαίδευση και τη ε, αγωγής του ε, πολίτη και η οποία καταλήγει σε παρόμοια μηνύματα όπως και η δική σας ε, ότι υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα εφαρμογής όλοι συμφωνούν ότι η ευαισθητοποίηση είναι σημαντική αλλά από την από την ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση υπάρχει ένα τεράστιο χάσμα. Ε, νομίζω λοιπόν ότι συμφωνούμε και πιστεύω ότι θα έχουμε μια πολύ σφαιρική εικόνα στο τέλος, ε, γιατί βλέπουμε από διαφορετικές οπτικές γωνίες ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ευχαριστήσω μία ακόμη φορά για την πολύτιμη εργασία σας. Με πολύ χαρά θα συνεργαστούμε με το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή Πολιτισμού ε, στο μέλλον και για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ Ακούσαμε και πολύ ενδιαφέρουσες ε, παρεμβάσεις. Ε, κύριε Φαγγελέ, έχετε τώρα τη δυνατότητα για πέντε λεπτά, αν μπορέσετε βέβαια το καταφέρετε αυτό, να απαντήσετε στα όσα ακούσατε. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τα θετικά σας σχόλια. Είμαστε πολύ ευτυχείς που ακούσαμε αυτά τα, σας τα σχόλια. Συνεργαστήκαμε με ειδικού από τις 28 χώρες και είχαμε πολύ αγαστή συνεργασία. Πραγματικά με σε πόσο αφοσιωμένοι είναι πολλοί ε, πανεπιστημιακοί ε, που εργάζονται σε αυτό το θέμα. Το θεωρούν όλοι εξαιρετικά σημαντικό. Γι' αυτό σας ευχαριστώ για τα θετικά σας ε, λόγια. Κάποιοι συζήτησαν την έννοια της ε, δημοκρατίας και της κουλτούρας της ανοχής. Όπως θα δείτε στην έκθεσή μας, δεν λέμε ότι η δημοκρατία και η ανοχή είναι συγκεκριμένες έννοιες. Έχουν ιδιαίτερο νόημα βεβαίως. Υπάρχουν κάποιες ιδέες για το τι σημαίνει επίσης ακριβώς η κάθε έννοια. Επίσης κάνουμε διάκριση ανάμεσα στις διάφορες έννοιες της δημοκρατίας και τις διάφορες ε, πετυχές εκφάνσεις της ανοχής. Λέμε ακόμα ότι η, η ανοχή είναι κατά την γνώμη μας πολύ αρνητική λέξη. Προτιμούμε άλλες λέξεις όπως ε, ε δέσμευση σεβασμού ε, κτλ. Υπάρχουν ένα σωρό άλλες έννοιες που σχετίζονται με την ανοχή. Και βεβαίω όλες αυτές οι έννοιες συνδέονται με την ελευθερία, την αξιοπροπία, την συμβίωση. Δεν λέμε δηλαδή ότι η παιδεία πρέπει να διδάξει αυτές τις αξίες, αλλά ότι ιδιαίτερα η παιδεία ε, μαθαίνει στα παιδιά και στους φοιτητές ε, που έχουν ένα διάλογο ε, τι ακριβώς σημαίνουν αυτές οι έννοιες και τι σημαίνουν και για τους ίδιους. Αυτό είναι το πολύ σημαντικό σε όλα τα επίπεδα. Επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μελών, επίπεδο σχολείων και τάξεις διδασκαλίας. Το σημαντικό είναι να γίνεται πολύς διάλογος για το τι σημαίνουν αυτές οι έννοιες. Είναι σημαντικό δηλαδή για ε, τα παιδιά και οι άνθρωποι να δέχονται αυτές τις αξίες γιατί είναι ε, θεμελιώδεις για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για την διδασκαλία των κοινών αξιών. Και όπως έλεγε και ο πρώτος ομιλητής, ε, συχνά έχουμε δει ότι η παιδεία μπορεί να είναι ουδέτερη ως προς τις αξίες. Ποτέ δεν γίνεται αυτό. Κάποιες φορές αμελούμε να μιλήσουμε για τις αξίες, αλλά δεν γίνεται να είναι ουδέτερη η παιδεία. Εγώ θα στήριζα ένα πιο θετικό, πιο δραστήριο, πιο ενεργό τρόπο για να σκεφτούν τις αξίες. Και έπειτα, τελική ερώτηση. Δεν έχουμε μια περιπτωσιολογική μελέτη για την Ιταλία, αλλά ο, τελικός, ο Ιταλός μας μας είπε κάποια πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για το γεγονός ότι η κυβέρνηση ζήτησε από τα σχολεία να συνεργαστούν με τις κοινότητες σε διάφορες ομάδες. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι μια από τις συστάσεις που αναφέρουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει πιο πολύ τοπική συνεργασία. Αυτό το εκτίμησα πάρα πολύ. πρέπει να προσπαθήσουμε λοιπόν εδώ να συμπεριλάβουμε τους ανθρώπους στη συζήτηση και κάναμε και κάποια έρευνα για τη διεθνοποίηση και την εθνικό προσανατολισμό. Η διεθνο... Η διεθνής προσανατολισμός αυξάνεται, καθώς και η προσανατολισμός προς την Ένωση. Ωστόσο, και η εθνική, ο εθνικός προσανατολισμός εξακολουθεί να είναι πολύ ισχυρός. Αλλά δεν είναι συχνά επικριτική στάση αν δούμε την ιστορικά τα πράγματα και στην Ολλανδία δεν είμαστε πολύ καλοί στο να βλέπουμε την ιστορία μας και τις κακές πλευρές της ιστορίας μας. Και αυτό λοιπόν θα πρέπει να το, να το συμπεριλάβουμε. Τώρα, από την Τσεχία είχαμε μια, ε, ε, ε, μια ερευνήτρια που είπε ότι πρέπει να προσθέσουμε συζητήσεις στις αίθουσες διδασκαλίες και γι' αυτό χειριζόμαστε ασφαλή σε αίθουσες διδασκαλίες αλλά και να στηρίξουμε τους δάσκαλους όταν αυτοί συζητούν θέματα πολύ πιο επίμαχα και αντιφατικά. Θα πρέπει να μπορούν να συζητήσουν τα πάντα. πρέπει να έχουμε δηλαδή πιο ανοιχτό κλίμα ως προς τις ιδεολογίες στο σχολείο. Καθώς και διαφορετικούς τρόπους διδασκαλές, όχι μόνο τους παραδοσιακούς, αλλά και πιο διαλογικού τύπου ε, διδασκαλία, να μάθουν οι ε, επιφοιτητές δηλαδή και οι μαθητές να είναι δημοκρατικοί, να μπορούν να συζητούν και να αποφασίζουν μαζί. Και φυσικά ήταν πολύ καλές και οι παρατηρήσεις της Κομισιόν ότι είναι αυτό η δική μας μελέτη σύμμορφη με άλλες, αλλά θέλω να αναφέρω μια μελέτη αυτό που λέμε gap in policy, δηλαδή κενά μέσα στην πολιτική, όχι ανάμεσα στις πολιτικές. Σε πολλές χώρες υπάρχουν πολύ ωραίοι γενικοί στόχοι, αλλά όταν φτάσουμε στα, στο διατάφτα και στις συγκεκριμένα μέτρα, εκεί κολλάει το πράγμα και υπάρχουν κενά. Θερμά σε ευχαριστίας και για τις απαντήσεις που μας δώσατε και για τις εκτιμήσεις σας. Νομίζω ότι και από τη συζήτηση φάνηκε ότι είναι πολύ σημαντική η μελέτη αυτή για τις ε, μελλοντικές μας εργασίες. Θα μας βοηθήσει πολύ και περιμένουμε και από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή μελλοντική συνεισφορά. Ελπίζουμε να μας υποστηρίξει γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα γιατί πρόκειται για το σύνολο των κοινωνιών. Θέλουμε να υπάρχει σύμπνοια στις ε, κοινωνίες μας. Και σίγουρα για να υπάρχει ειρήνη και ειρηνική συμβίωση κοινωνίας θα πρέπει να νιώθουν όλοι οι πολίτες ότι ανήκουν ε, στην κοινωνία, ανήκουν ε, στη χώρα. Μιλήσατε για αυτά τα gap, για αυτά τα κενά θα τα συζητήσουμε, πρέπει να τα συζητήσουμε κατεπηγόντως τα επόμενα χρόνια ώστε στο μέλλον να μην έχουμε τόσα άτομα τα οποία νιώθουν ε, αφημένα στη μοίρα τους, ε, αλλά αντίθετα να βοηθήσουμε όλα αυτά τα άτομα να ταυτιστούν με την κοινωνία στην οποία ζουν. για να καταπολεμηθούν και ακραία φαινόμενα. Πιστεύω ότι Θα πρέπει τα παιδιά μας να μπορούν να, να ε, διαλέγονται, να συζητούν, να καταλάβουν τι θα πει δημοκρατία και ποιες αξίες συνδέονται άρρηκτα με τη δημοκρατία. Τέτοια μέτρα πρέπει να προωθήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που σας εδώ σήμερα. können nahtlos weitermachen. Μπορούμε να συνεχίσουμε χωρίς διακοπή. Μόλις έφτασε και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επόμενο θέμα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε λοιπόν και ερχόμαστε στο 7 ανταλλαγή απόψε με την Επιτροπή Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Έτσι Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να συζητήσουμε είναι η υλοποίηση Θέλω να ευχαριστήσω πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που έδειξε προθυμία να έρθει εδώ σήμερα για να μας ενημερώσει, να απαντήσει στις ερωτήσεις της Επιτροπής μας και δεν νομίζω ότι προδίδω και κανένα μυστικό άμα σας πω ότι για την Επιτροπή μας ε, το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς είναι κάτι που μας είναι ιδιαίτερος προσφυλές, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί έχει να κάνει και με την σημασία που αποδίδουμε εμείς στην ε, πολιτιστική κληρονομιά, είτε είναι ηλική είτε άειλη, αλλά σχετίζεται επίσης και με το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν αυτό που με πάρα πολύ μεγάλη έμφαση ε, πάλεψε να υπάρχει αυτό το έτος και γι' αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να συνεισφέρουμε στην επιτυχία αυτού του έτους. Και επομένως θέλουμε να δούμε ότι και αυτή τη χρονιά θα στεφθεί με επιτυχία. Ε, το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής ε, Κληρονομιάς. Ξέρω ότι υπάρχουν προετοιμασίες στο πλαίσιο της αρμόδιας γενικής διεύθυνσης και θα ήθελα και από δικής μας πλευράς ε, να σας διαβεβαιώσουμε ότι πρέπει να έχετε, να συνειδητοποιήσετε ότι έχετε στο πρόσωπό μας πιστούς ε, παρότι μπορεί βέβαια κάποιες φορές να ασκούμε την κριτική μας. Σε ό,τι αφορά τώρα τα θέματα τα οποία μας ενδιαφέρουν, το ένα είναι η συμμετοχή του Κοινοβουλίου στη συζητήση με τους εμπλεκομένους ε, και τις προθεσμίες ε, για τις συνεντήσεις των εθνικών συντονιστών. Για αυτά τα δύο θέματα, με γραπτή διαδικασία, ε, ανταλλάξαμε τις απόψεις και υπήρξε η επιστολή Ναύρατσιτς ότι πράγματι θα συμμετέχουμε σε αυτές τις διαβουλεύσεις με τους stakeholders. Έχουν ρυθμιστεί και τα σχετικά με την ε, συνάντηση των εθνικών συντονιστών. Απλά πρέπει να δούμε τι ημερομηνίε για να μην συμπίπτουν με συνεδριά της δικής μας Επιτροπής. θα τα ξεκαθαρίσουμε όμως, δεν υπάρχει πρόβλημα. Επίσης, στην επιστολή ε, σας είχαμε ζητήσει να μην μας πείτε μόνο ε, τι θα γίνει με το επόμενο έτος ε, και πώς θα, θα πανεθούν τα κονδύλια και για φέτος τι θα γίνει που έχουμε ένα εκατομμύριο ευρώ. Μπορεί να μην είναι πάρα πολλά, παρόλα αυτά όμως μπορούν αυτά τα χρήματα να αξιοποιηθούν καταλήλως ώστε να συνεισφέρουν ε, στην ε, βελτίωση των εκδηλώσεων για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στην τελευταία συνεδρία των συντονιστών διαπιστώσαμε ότι ιδίως ό,τι αφορά τον προϋπολογισμό. Υπάρχουν κάποια ζητήματα σε ό,τι αφορά την κραμιστον των κονδύλων και θα ήθελα ήδη να σας ενημερώσω για τις ε, ερωτήσεις μας. Σε ό,τι αφορά τη συνάντηση των εθνικών συντονιστών, υπάρχει το ποστό 200.000 δεν μας ικανοποιεί ακριβώς, κύριε Μαγνιέ. Γιατί ε, κοστίζει τόσο πολύ αυτή η συνάντηση των εθνικών συντονιστών. Μήπως να τα διαθέτατε καλύτερα κάπου αλλού αυτά τα χρήματα. Αυτή είναι μια ερώτηση που μας δημιουργήθηκε ε, στη συνεδρία των συντονιστών, αλλά φαντάζομαι ότι θα μας δώσετε ικανοποιητικές απαντήσεις ε, στη συνέχεια. Θα σας δώσω λοιπόν κύριε Μανιέ το λόγο για να μας ενημερώσετε για το πώς έχουν τα πράγματα. Θα έλεγα 10 λεπτά να διαρκέσει η παρουσίασή σας, οπότε να μπορέσουμε μετά, αν υπάρχουν ανοιχτά θέματα, να τα ξεκαθαρίσουμε στο διάλογο που θα το ακολουθεί. Σας ευχαριστώ και πάλι που είστε εδώ, έχετε το λόγο. Donc je vais essayer pendant les 10 euh, minutes. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω στη διάρκεια των 10 λεπτών που μου δώσατε να σας παρουσιάσω τι έχουμε ήδη κάνει από την έναρξη ισχύω της νομικής βάσης για το πολιτιστικό έτος, δηλαδή μετά το τέλος ε, Απριλίου. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την πρόσκληση για να έρθω στην Επιτροπή Πολιτισμού και να σας πω ότι είμαστε έτοιμοι να ερχόμαστε τακτικά για να σας ενημερώνουμε για το τι έχουμε κάνει και για την κατάσταση πρόοδου ε, της, των ε, προετοιμασιών για το έτος. Θέλω να αναφερθώ στο θέμα της διακυβέρνησης και της εταιρικότητας που είναι σημαντικά για μια τέτοια πολιτιστική χρονιά. Έχουμε λοιπόν ε, φτιάξει τις δομές που θα μας επιτρέψουν να χειριστούμε ε, να διαχειριστούμε το έτος και έχουμε κάνει μια συνεδρίαση με τους 28 εθνικούς συντονιστές, των οποίων ο ρόλος θα είναι φυσικά εξαιρετικά σημαντικό σε επίπεδο και των μελών. Επίσης, επιλέξαμε 35 stakeholders ε, ε, ενδιαφερόμενους φορείς της κοινωνίας των πολιτών για να αποτελέσουν μέρος της Επιτροπής που μας βοηθεί, βοηθάει για τη διοργάνωση του έτους και διοργανώσαμε και την πρώτη συνεδρίαση αυτής της Επιτροπής. Προγραμματίσαμε και άλλες συνεδριάσεις αυτών των δύο Επιτροπών και παντώ, κυρία Πρόεδρε, αμέσω το ερώτημά σα είναι για, να διοργανώ... για τη διοργάνωση αυτών των έξι ε, συνεδριάσεων που θα χρησιμοποιήσουμε τα 200.000 ευρώ. Δεν πρόκειται για μία συνεδρίαση, αλλά για έξι 36 τον αριθμό. Κάθε φορά ε, συγκεντρώνονται 30-35 συμμετέχοντες. Θα δουλέψουμε λοιπόν κατά προτεραιότητα με τις υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας που παίζει σε απέξ ρόλο στην ε, εκστρατεία επικοινωνίας για αυτό το έτος και έχουμε έρθει σε επαφή με ολόκληρη τη Γενική Διεύθυνση που έχουν δραστηριότητε ε, που έχουν να κάνουν με το πολιτισμό, DG έρευνα, DG home, DG περιβάλλον, DG ανάπτυξη έχουν όλες αυτές οι γενικές διευθύνσεις δράσεις που, ετοιμάζονται ή που τρέχουν, που συνδέονται οικονομικά με το ευρωπαϊκό έτος και φυσικά αυτές οι δράσεις θα αποτελέσουν και τμήμα ε, των δράσεων για αυτό το έτος. Στη δική μας γενική διεύθυνση παρουσιάσαμε το ευρωπαϊκό έτος στους εθνικούς ε, ε, εκπροσώπους έρασμο ε, Συν για να του επιτρέψουμε να συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό Έτο, γιατί ξέρετε ότι η νεότηση και η παιδεία είναι, παίζουν σημαντικό ρόλο. Μέσα από την επικοινωνία λοιπόν και τα ανακοινοθέντα μας θα ενημερώσουμε όλες τις αντιπροσωπείες στα κράτη-μέλη για να τις καλέσουμε να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους για αυτό το χρόνο και επίσης θα συναντηθούμε με δύο θεσμούς που παίζουν σημαντικό ρόλο, την Επιτροπή των Περιφερειών και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ώστε να δούμε ποια θα μπορούσε να είναι η δική του συμβολή στην, ε, στο και πέρα από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα συνεδριάσαμε με πολυάριθμους ε, διεθνείς οργανισμούς όπως η UNESCO, η, το Συμβούλιο της Ευρώπης, ε, η ΚΡΟΜ, η ΚΟΜΟΣ, όλα, όλοι οι διεθνείς οργανισμοί που ασχολούνται με την κληρονομιά και Έχουμε έρθει σε επαφή με άλλους οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή και το Google Cultural Institute, ε, το πολιτιστικό Ινστιτούτο του Google που έχει αναπτύξει ένα project που θα μπορούσε να είναι καλό για την κληρονομιά. Τώρα, ε, προπολογισμό. Να αρχίσω με το 2017. Για το 2017 έχουμε ένα εκατομμύριο ευρώ, το οποίο χορηγήθηκε από το Κοινοβούλιο και μάλιστα θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι για αυτό το κονδύλι, για τη συγκεκριμένη αυτή δέσμευση που μας επιτρέπει να προετοιμάσουμε το ευρωπαϊκό έτος. Αυτός ο προπολογισμό βοηθά στην προετοιμασία του 2018 και τα, οι δαπάνε κατανέμονται σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη με 260.000 ευρώ είναι ένα ευρωβαρόμετρο που θα μας επιτρέψει να μετρήσουμε την αντίληψη των πολιτών για την πολιτιστική κληρονομιά. Αυτό το μέσο θα είναι εξαιρετικά χρήσιμο στο να κινητοποιήσουμε τον τύπο και τα ΜΜΕ είναι η εμπειρία από όλα τα ευρωπαϊκά έτη ώστε τύπος ε, να ενδιαφέρεται για, ε, ε, για το έτος πολιτιστικής οικονομίας. Κάθε χρόνο γίνεται ένα τέτοιο ευρωβαρόμετρο. Δεύτερη κατηγορία δαπάνης είναι η επικοινωνία. 500.000 ευρώ. Έχουμε μια σύμβαση με έναν εξωτερικό συνεργάτη για να προετοιμάσει μια οπτική ταυτότητα, σαφή μηνύματα, καθώς και μια ταινία. Να τονίσω ότι οι εθνικοί συντονιστέ ε, επιτοπλίστων δήλωσαν ότι θέλουν να χρησιμοποιήσουν τη δικό μα σήμα, αυτό και τα δικά μα μηνύματα κλειδιά, ώστε να υπάρχει μια συνοχή στο μήνυμα. Και αυτό είναι εξαιρετικά θετικό, γιατί εγγυάται μια ε, επικοινωνία συνεπή και παρόμοια για όλο την, ε, το, το πολιτιστικό έτος. Ε, έχουμε φτιάξει και ένα site γιατί όπως γνωρίζετε είναι απαραίτητο αυτό. Ε, ελπίζουμε να έχουμε και ένα λάβαρο πάνω στο Μπερλεμό ε, για να είναι ορατή η, χρονιά, η πολιτιστική χρονιά για όλους στο δημόσιο χώρο και επίσης θα ενημερώσουμε τα σχολεία ε, σε όλες τις γλώσσες έχουμε φυλάδια και έχουμε διοργανώσει παιχνίδια και ένα διαχωνισμό για να ε, προσελκύσουμε τους νέους που είναι ο κατεξοχήν στόχος αυτής της χρονιάς. Ε, και όλα αυτά ήδη θα υπάρχουν το 17 ώστε να υπάρχουν να είναι διαθέσιμα όταν θα ξεκινήσει η χρονιά. Αυτός ο προπολογισμό είναι αρκετά σημαντικός να συγκρίνουμε το Ευρωπαϊκό Έτος της Ανάπτυξης που έγινε το 2015 με 11 εκατομμύρια ευρώ περίπου 3,5 εκατομμύρια ευρώ ήταν τότε το κονδύλι για την επικοινωνία, πολύ μεγαλύτερο δηλαδή. Πιστεύουμε πως έτσι γίνονται πιο ουσιαστικές δράσεις και θα επανέλθω σε αυτές σε λίγο. Και τέλος ε, φέτος το 2017 έχουμε 200.000 ευρώ για τις συνεδριάσεις των εθνικών συντονιστών και των φορέων της κοινωνίας των πολιτών, δηλαδή 6 συνεδριάσεις στο σύνολο για το 2017 είναι αυτό απαραίτητο, γιατί όπω έλεγα η χρονιά αυτή είναι μια διαδικασία που πρέπει να συμμετέχουν όλοι. Οι συνεδριάσει αυτέ έχουν ήδη προγραμματιστεί και είναι εξαιρετικά χρήσιμε για την προετοιμασία του 2018. Εάν κάνετε τη σούμα, μένουν 40.000 ευρώ που θα τις κρατήσουμε για πρόβλεπτες δαπάνες. Να στιγμή δεν χρειάστηκε να τα χρησιμοποιήσουμε να επιμείνω για το ότι άλλες δαπάνες για το ευρωπαϊκό έτος θα αναλυθούν από άλλες γραμμές, ας πούμε φόρουμ πολιτισμού που θα γίνει φέτος το Δεκέμβριο στο Μιλάνο και εκεί αυτό θα χρηματοδοτηθεί από άλλο κονδύλι. Επίσης χρησιμοποιούμε τον προπολογισμό της δικής μας Γενικής Διεύθυνσης για διάφορες, εκπομπές, για διάφορες αποστολές και ενίσχυση του προσωπικού που χρειαζόμαστε. για την προετοιμασία. Όσον αφορά τις ίδιες τις δραστηριότητες, να σας πω σύντομα, έχουμε τρία επίπεδα που θα είναι τα πιο ενεργά. Έχουμε το ευρωπαϊκό επίπεδο που θα γίνουν δράσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να ε, δείξουμε διάφορα θέματα και να ε, προωθήσουμε διάφορα project που ε, έχουν ευρωπαϊκή διπροσθεμένη αξία. Έχουμε 10 ε, ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, τις θα διαχειριστούμε άμεσα εμείς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. και που θα επιτρέψουν να, συνεχιστούν, να συνεχιστεί η συζήτηση πέρα από το 2018. Θα είναι η κληρονομιά που θα αφήσει το έτος ώστε να προκύψουν και πιο πολιτικέ συζητήσει για αυτά τα θέματα. Δεύτερο επίπεδο δράση, διακρατική συνεργασία, γιατί είναι σημαντικό όλοι οι φορεί που ασχολούνται με την κληρονομιά να συνεργάζονται διασυνοριακά, διακρατικά και έχουμε την πρόθεση να ξεκινήσουμε το Σεπτέμβριο μια προκήρυξη ενδιαφέροντος ε, για προτάσεις, ε, για επιδοτήσεις ε, στον τομέα της ε, κληρονομιάς και έχουμε κρατήσει μεγάλο κομμάτι της χρηματοδότησής μας 20 με 25 project προγραμματίζουμε να έχουμε και το τρίτο επίπεδο δράσης θα είναι το εθνικό βεβαίως όπου αυτό εξαρτάται από τους εθνικούς συντονιστές στους οποίους θα στείλουμε ένα πίνακα να συμπληρώσουν για να έχουμε μια ήδη πρώτη ιδέα για το τι δραστηριότητες σκοπεύουν να οργανώσουν. Να τονίσω ακόμα ότι έχουμε οργανώσει αυτή τη βδομάδα μια συνεδρίαση υπευθύνων για τις Ευρωπαϊκές ημέρες ε, ε, κληρονομιά για να δώσουμε μια όθηση στο πρόγραμμα αυτό που αγγίζει μια τριανταριά εκατομμύρια πολίτες κάθε χρόνο και το οποίο η ευρωπαϊκή διάσταση θα πρέπει να προωθηθεί περισσότερο. Το 2018 λοιπόν οι ευρωπαϊκές ημέρες κληρονομιάς θα πρέπει να είναι πιο ορατές και να έχουν πιο ξεκάθαρα ευρωπαϊκή διάσταση. Να τονίσω ε, επίσης ότι χρησιμοποιούμε διάφορα προγράμματα σε επίπεδο περιφερειών και πόλεων. Έχουμε ήδη κάποιες επαφές, ε, μέγα ενδιαφέρον έχουν δείξει πόλεις και περιφέρειες ε, και θέλουμε να συνεργαστούμε σε αυτό το επίπεδο με τα δίκτυα των πόλεων, όπως το EuroCities ή ενώσεις περιφερειών ή πόλεων. Επίσης ε, θα ξεκινήσουμε τη χρονιά με δύο ευκαιρίες. Πρώτον ε, το φόρουμ του πολιτισμού που θα γίνει στο Μιλάνο το Δεκέμβριο και επίσης ε, υπάρχει μια εκδήλωση γκαλά που θα οργανωθεί από την Βουλγαρική Προεδρία στη Σόφια στις 11 και 12 Ιανουαρίου κατά την συνήθη παραδοσιακή συνάντηση μεταξύ της Προεδρίας και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πρόκειται για δύο ευκαιρίες που θα είναι πολύ καλές για να κάνουμε μια ε, δημοσίευση ή μια προώθηση ε, της, ε, του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Μανιέ. Λοιπόν, για να δούμε ποιοι είναι στον κατάλογο. Πρώτη είναι η κυρία Σιλβία Κώστα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Η παρουσίαση που μας κάνατε έχει λάβει υπόψη πολλά από τα αιτήματα που υπευλήθησαν την πρώτη συνάντηση στις 25 Απριλίου από τα κράτη-μέλη και από το Κοινοβούλιο και ας πούμε, να ξεκαθαρίσουμε καλύτερα πώς ε, θα δαπανηθούν ε, οι πόροι του 2017 για την επικοινωνία και να είναι μια επικοινωνία επικοινωνική στρατηγική που θα ε, προσελκύσει περισσότερο τους νέους, τους stakeholder, τις περιφέρειες και όλους. Ε, μιλήσατε όχι μόνο για το λόγο και την ταινία που έχει γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και διάφορους τρόπους πέρα από το web, για να προχωρήσει από τα κάτω προς τα πάνω. Μια δημιουργικότητα νεανική που να αισθανθεί ότι συμμετέχει και αυτή. Πολύ σημαντικό αυτό. Έπειτα έχουμε το φόρουμ του Μιλάνο. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό το Δεκέμβριο, αλλά είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πότε θα έχει ετοιμαστεί το υλικό. Το λόγο, το σήμα, όλα, το, το, kit όλο. Για να, οι θετικοί συντονιστέ είναι έτοιμοι για να συμμετέχουν. Οι δέκα βασικέ πρωτοβουλίε τώρα. Ένα από τα αιτήματα που έχουμε κάνει είναι ε, ε, το έτος να μην τελειώσει με το τέλος του 18, αλλά να ξεκινήσουν κάποια μεγάλα θέματα που αφορούν ε, οριζόντια την, την κληρονομιά και που θα μπορούσαν να γίνουν ε, και οι flag initiatives. Εσείς είπατε ότι θα προταθούν όλα αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θέλω να ξέρω, το Κοινοβούλιο θα συμμετέχει σε αυτή την ομάδα συντονιστή, τη συντονιστική, αν υπάρχει ήδη κάποιο διάλογο και σε τι επίπεδο με τα κράτη-μέλη. Να καταλάβω αν θα υπάρξει μια κατανομή για τα θέματα ε, το ποια θα είναι τα θέματα που θέλουν να εξεταστούν, με ποια και γεωγραφική ισορροπία. Κάτι ακόμα που ζήτησε και είναι καλό που αρχίσατε τη διαβούλευση με αυτό το θέμα, δηλαδή ε, ε, ο και Περιφερειακή Επιτροπή, Επιτροπή των Περιφερειών μάλλον, Ομάδα εργασία τώρα συντονισμού και Επιτροπή των διαφερόμενων φορέων, των συμμετεχόντων φορέων. Νομίζω ότι στι 6 Σεπτεμβρίου έχετε προβλέψει μια σύνδεση μεταξύ των δύο αυτών ε, επιτροπών. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για τον διαγωνισμό, νομίζω 5.000 ευρώ θα πρέπει να μπουν στον διαγωνισμό ε, Δημιουργική Ευρώπη και από την άποψη των πρωτοβουλειών, νομίζω πως κάποιες χώρες έχουν ήδη κατά κάποιο τρόπο εντοπίσει δραστηριότητες, προτείνει δραστηριότητες και θα πρέπει να δείτε με τους εθνικούς συντονιστές πόσο και ποιοι φορείς ε, συμμετέχουν, να μην είναι μονοκρατικοί φορείς και κάτι ακόμα το οποίο θα μας αφορά εμάς είναι η συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων. Αυτό είναι δική μας δουλειά, γιατί πρέπει να υπάρξει συνεργασία. Πολλές χώρες δεν ξέρουν πολλά ε, όσον αφορά τους ε, θεσμούς. Κάτι ακόμα που έχουμε ρωτήσει. Τα άλλα προγράμματα, πώς οι άλλε SDG, πώ συνεργάζονται όσον αφορά τα προγράμματα που πρέπει να αφιερωθούν ε, στην πολιτιστική κληρονομιά. Είναι αυτό ένα, ερώτημα που είχαμε κάνει. Ξέρουμε ότι υπήρξαν πολλές κινήσεις, αλλά να μας πείτε λίγο αναλυτικότερα τι έγινε. Τώρα, πολιτιστική διπλωματία. Την επόμενη εβδομάδα ε, εγκρίνουμε το κείμενο. Ξέρω ότι από πλευρά των διαφόρων DG, DEFCO και άλλων ε, ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν συγκεκριμένα με κάποιε δράσει και project ήδη από το 2018, συνδυάζοντα και το ευρωπαϊκό Έτο. Γιατί, Γιατί η διάσταση προ τι τρίτε χώρε για μα είναι πολύ σημαντικό. Ποιε θα είναι οι τρίτε χώρε προ τι οποίε ε, θέλετε να στραφείτε και να συμμετέχουν. Είναι εκείνε τη ε, Δημιουργική Ευρώπη να ξεκαθαρίσουμε καλύτερα αυτή την πτυχή. Γιατί δεν είναι σαφέ ποιε θα είναι οι χώρε που θα μπορέσουν ανοιχτά να συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σόντροβα. Ευχαριστώ στα γαλλικά. Θέλω να ευχαριστώ θερμά τον κύριο Μανιέ. Είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω στην πρώτη συνάντηση και μπορώ να σας ε, μεταφέρω ότι πραγματικά υπήρχε μεγάλη προσέλευση, εκπροσωπήθηκαν όλες οι χώρες, υπήρχαν εμπειρογνώμονες, μεγάλο ενδιαφέρον, πολλές οι ερωτήσεις, πολλές οι προτάσεις για τη βελτίωση του προγράμματος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω επίσης που και τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήμασταν εκεί ως παρατηρητές και διαπιστώσαμε όλες αυτές τις δραστηριότητες από κοντά. Γιατί αυτό μας δίνει τη δυνατότητα ακόμη για καλύτερη συνεργασία. Ευχαριστώ λοιπόν γι' αυτό. Έχω την ίδια ερώτηση με τη συνάδελφό μου τη Σίλβια Κώστα. Πριν ένα μήνα μιλήσαμε για το λογότυπο, για την, κοινωνική, συγγνώμη, για την κοινή ταυτότητα και είπατε είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το προετοιμάσουμε. Πότε να το περιμένουμε. Έστω μήνα δώστε μας, έτσι, με κάπως μεγαλύτερη ακρίβεια. Αυτή την ταυτότητα ή αυτό το εγχειρίδιο, που πότε θα το έχετε έτοιμο. Ένα άλλο ερώτημα για την ε, εγγενίαση. Το έτος δεν ξέρω, στο Βερολίνο ίσως θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να συμμετέχουμε στο, στην εκδήλωση αυτή. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο χρονοδιάγραμμα για την ε, γενίαση του έτους. Στο Βερολίνο. Α, όχι στο Βερολίνο, στο Μιλάνο. Α, στο Μιλάνο. Θα ήθελα να μου πείτε ακριβώς ε, τις αν ε, μπορείτε. Για να το γράψουμε στις ατζέντες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Σαμπίνε Φερχάιν. Ένα σημείο συγκεκριμένα θέλω να σχολιάσω. Πράγματι, θέλουμε να υπάρχει βιώσιμη επιτυχία ε, στο ευρωπαϊκό έτος. Έχουμε φτάσει στη μέσα του έτους, μετά έχουμε καλοκαίρι και έχει μείνει μισός χρόνος. Ε, πολύ λίγος δηλαδή ε, το μόνο που έχω ε, είναι ότι φαίνεται να μην έχουμε προχωρήσει πολύ σε ό,τι αφορά το συντονισμό και στη διάρθρωση του έτους. Το ερώτημα είναι λοιπόν, με αυτά τα μέσα που έχουμε, πώς μπορούμε να προχωρήσουμε ε, και να πιέσουμε πιο ισχυρά, πιο έντονα μετά το καλοκαίρι, μετά τη στερινές διακοπές, να μην είναι lame duck, Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Χέλγκα Τρουπέλ, ναι. Και εγώ θα ήθελα να σχολιάσω αυτό που είπε η Σαμπίν. Μέχρι στιγμή, τουλάχιστον και όταν μιλάω στη Γερμανία με κάποιου από του εμπλεκόμενου φορεί, λένε ότι δεν νιώθουν ότι του έχουν ενημερώσει. Ούτε καν έχουν καταλάβει ότι έρχεται αυτή η χρονιά, αυτό το ευρωπαϊκό έτο και σε επίπεδο των εξωτερικών ε, που λένε ότι δουλεύουν, αλλά αν μιλήσει κανεί με φόρου μουσείων και άλλου πολιτιστικού φορεί σε τοπικό επίπεδο, διαπιστώνει ξεκάθαρα ότι δεν ε, έχουν καταλάβει τι θα συμβεί ακριβώ. Άρα, τι κάνετε εσεί για να βελτιώσετε ε, τι επαφέ και αν υπάρξει αυτή η επαφή, εμεί οι απλοί πολίτε και άλλοι, όχι μόνο εμεί, πώ θα δουν ε, τι περιλαμβάνεται σε αυτές τις ε, εκδηλώσεις. Το λόγο, η ορατότητα, η προβολή, μιλήστε για ένα βίντεο κτλ. Αλλά πώς θα ενημερώσετε τη βάση, την τοπική κοινωνία. Πώς θα τους ενημερώσετε, ποιες δραστηριότητες περιλαμβάνει το ευρωπαϊκό έτος. Δεν υπάρχει διαφάνεια, κατά μέχρι στιγμής. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Μια στρατηγική bottom-up από κάτω προς τα πάνω μπορεί να λειτουργήσει μόνο εάν η βάση ξέρει τι γίνεται ε, από στην κορυφή. Αν όχι, εγώ έχω μια ερώτηση, αν μπορείτε να μας πείτε λίγο παραπάνω για αυτές τις 10 εμβληματικές πρωτοβουλίες, αυτά τα 10 project. Αν μπορούμε να έχουμε λίγο περισσότερες πληροφορίες. Και τώρα μπορώ να σας ξαναδώσω το λόγο για να μας απαντήσετε σε αυτά τα ερώτηματα, κύριε Μανιέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κράτησα τη δική σας ερώτηση για το τέλος και θα απαντήσω πρώτα στις πρώτες ερωτήσεις. τα εργαλεία επικοινωνία. Είμαστε πολύ απογοητευμένοι που δεν τα έχουμε ήδη στη διάθεσή μα. Θα θέλαμε να τα έχουμε στη διάθεσή μα. Τα περιμένουμε όμω ε, ο ε, υπεύθυνο του έργου πρέπει να τα επεξεργαστεί και να τα επαληθεύσει. Ελπίζουμε πάντως αρχές Σεπτεμβρίου να μπορούμε να τα έχουμε στη διάθεσή μας. Θα ενημερώσουμε τα κράτη-μέλη, ε, τους έχουμε πει ήδη δηλαδή ότι θα είναι διαθέσιμα τότε ό,τι και να γίνει. Μπορώ να δεσμευθώ ότι θα συμβεί αυτό. Τουλάχιστον προς αυτή την κατεύθυνση εργαζόμαστε. Είναι γεγονός ότι κάποια κράτη-μέλη έχουν αρχίσει πολύ ενεργά ε, να ε, δουλεύουν ήδη. Η Γερμανία, για παράδειγμα, έχει ήδη μία ταυτότητα ε, οπτική ε, είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Έχει ξεκινήσει διάφορες εκδηλώσεις επίσης. Κάποια άλλα κράτη-μέλη έχουν αρχίσει κάποιες εθνικές εκδηλώσεις για να υπάρξει αυτή η συνειδητοποίηση σε επίπεδο πολιτιστικών ε, φορέων ε, της περιοχής. Εμείς πιστεύουμε ότι η κρίσιμη χρονική στιγμή θα είναι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Ε, τότε θα αρχίσει να εκδηλώνεται το ενδιαφέρον, ε, τότε θα επισπεύσουμε τις εργασίες μας, θα έχουμε όλες αυτές τις ταυτότητες, τα λογότυπα στη διάθεσή μας και θα είναι για μας πολύ ευκολότερο να παρουσιάσουμε κάτι το συγκεκριμένο. Η συνεργασία με τις άλλες γενικές διευθύνσεις γίνεται με πολύ ομαλό τρόπο, πολύ καλύτερα από ό,τι περιμέναμε. Δεν είναι δικό μας σε αυτό το εγχείρημα, είναι ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα και όλες οι δραστηριότητες όλων των γενικών διευθύνσεων που ε, συμμετέχουν, όπω η Γενική Διεύθυνση έρευνα, α πούμε, είναι πάρα πολύ ενθουσιώδης. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ χρήσιμα. Ανάπτυξης, ε, Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης. Έχουμε πάρα πολύ θετική ανταπόκριση και πιστεύουμε ότι του χρόνου θα δείτε πολλούς επιτρόπους να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του Ευρωπαϊκού Έτους. Η πολιτιστική διπλωματία φυσικά είναι μια σημαντική διάσταση. Θα συνεργαστούμε με τις ε, αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως ε, στις 2 η ώρα του απόγευμα έχουμε στον Περλεμόν μια ενημερωτική συνεδρίαση με τις τρίτες χώρες, όλες οι τρίτες χώρες που συμμετέχουν ε, στη Δημιουργική Ευρώπη και θα δούμε σε ποιο βαθμό θέλουν και εκείνε να συμμετάσχουν. Ήμουν στο Στρασβούργο, στο Συμβούλιο της Ευρώπης πριν από ένα μήνα και είδα Διαπίστωσα ότι όλα τα μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης ενδιαφέρονται πολύ να συμμετέχουν σε, αυτήν την, ε, σε αυτό το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Προφανώς ο προπολογισμό ε, ε, προέρχεται από ε, τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε αυτά ε, αποσκοπεί παρόλα αυτά κάποιες χώρες, η Ελβετία για παράδειγμα μας είπε ότι ενδιαφέρεται να δρομολογήσει πολλές δραστηριότητες, κάτι το οποίο βέβαια θα συνεισφέρει στην ορατότητα της, του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Τώρα, πότε θα εγγενιάσουμε τη χρονιά. Ε, στο πολιτιστικό φόρουμ που γίνεται κάθε δύο χρόνια, αυτή τη φορά ένα τμήμα θα είναι ε, τα, η επίσημη έναρξη του Ευρωπαϊκού έτους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίως θα ε, συμμετέχει σε, αυτό το, ε, σε αυτή την εκδήλωση στο υψηλότερο δυνατό ε, επίπεδο. Έχουμε ήδη πει ε, στην κυρία Καμερβέρ τις ημερομηνίε ώστε να μπορέσει να τις λάβει υπόψη στην, στο πρόγραμμά της. γνωρίζουμε ότι έχουμε πραγματικά μπροστά μας έναν αγώνα δρόμου να δώσουμε. Πρέπει να κάνουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε για τη ε, νομική ε, βάση. Καταφέραμε να την εγκρίνουμε, λύσαμε πολλά διοικητικά προβλήματα και προσπαθούμε να πάμε όσο το δυνατόν ε, ταχύτερα. Γι' αυτό ακριβώς, κυρία Πρόεδρε, αναλάβαμε την ευθύνη οργάνωσης της πρώτης συνάντησης εθνικών συντονιστών δύο μέρες μετά την έναρξη ισχύω της νομικής βάσης. Νομίζω ότι ήταν συνετό αυτό. Ε, μας λείπουν κάποιοι μήνες για να είμαστε απολύτως ε, άνετοι με το χρονοδιάγραμμα. Πρέπει να είμαστε γρήγοροι, πρέπει και εμείς να κάνουμε προσπάθειες από πλευράς μας και αυτό κάνουμε. Όσον αφορά τα 10 ευρωπαϊκά ε, προγράμματα, αν έχουμε λίγο χρόνο, μπορούμε να σας κάνουμε μία, μία σύντομη παρουσίαση, αλλά μας χρειάζονται 10 λεπτάκια. Αλλιώς μπορούμε να κάνουμε την παρουσίαση και άλλη φορά. Εντάξει, 10 λεπτά. Να παρακαλέσω τότε την Κατρίνα να κάνει μια γρήγορη παρουσίαση. Θα εξηγήσω με τα θέματα το πώς προχωρούμε. Αλλά αν θέλετε πιο αναλυτική, μια άλλη φορά μπορούμε να σας πούμε πιο πολλά. Ναι, λοιπόν, ευχαριστώ Μισελ. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν εγώ αυτά τα 10 τα εμβληματικά project για το επόμενο έτος πολιτιστικής κληρονομιάς, αλλά πρώτα να αναφερθώ στο ερώτημα της κυρίας Τρούπελ, ε, που λέει ότι πρέπει να γίνει γνωστό το ευρωπαϊκό το σωστό να το περισσότερο στους πολίτες μας. Αυτός είναι ο στόχος μας Προφανώ γι' αυτό και ε, έχουμε το... Έχουμε, θέλουμε τη βοήθεια των λεγόμενων multipliers. Έχουμε πάνω από 300, 350 οργανώσεις που εξειδικεύονται στον τομέα του πολιτισμού και ενημερώνονται σε τακτά διαστήματα για τα θέματα του Ευρωπαϊκού έτους. Έχουμε όμως και πολλούς άλλους, πολλά σημεία επαφής ε, από τις αντιπροσωπείς της Κομισιόν, τις αντιπροσωπείς του Κοινοβουλίου Ελπίζουμε, έχουμε τις αντιπροσωπείς της τρίτες χώρες, έχουμε τα desk Creative Europe. στα εθνικέ υπηρεσίε του Erasmus Plus έχουμε εκείνη επίσης κάνει μια παρουσίαση, οπότε ελπίζουμε ότι έτσι θα μπορέσει να μεταφερθεί ε, πολύ πιο γρήγορα από ό,τι μπορούμε να κάνουμε εδώ στις Βρυξέλλες ε, ε, ό,τι έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό Έτο, Έχουμε μιλήσει με την ΕΟΚΕ και με την Επιτροπή των Περιφέρειων για να μα βοηθήσουν και αυτοί να μεταφέρουν τι πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Έτος στου συνομιλητέ του και ελπίζουμε να έχουμε και μία σε βάθος συζήτηση με τα τμήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που σίγουρα θα μας βοηθήσουν επίσης. Και τώρα έρχομαι στις 10 εμβληματικέ πρωτοβουλίες. Γιατί οι συγκεκριμένες πρώτα απ' όλα. Διότι θεωρούμε ότι πράγματι, εκτός της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, για τους πολιτιστικούς φορείς μέσω του Creative Europe, που είναι σίγουρα ένα σημαντικό πρόγραμμα, αλλά ουσιαστικά δεν ε, Μα επιτρέπει να διοχετεύσουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε, δεν θα ξέρουμε το πρώτο τι θα γίνει, για να συμπληρώσουμε αυτή την προσέγγιση, θέλουμε να έχουμε αυτά τα 10 project. Εμεί τα, τα ε, προετοιμάζουμε σε συνεργασία φυσικά με τα κράτη-μέλη, με σημαντικού εταίρες όπως η UNESCO και το Συμβούλιο τη Ευρώπη. Έτσι αποκρισταλώνεται η συνεργασία μας με τους διεθνείς οργανισμούς. Ξέρετε ότι κοινοβούλοι και κράτη-μέλη βοήθησαν και μάλλον επέμειναν να είναι εταίροι μας και είναι υποχρέωσή μας με βάση τη νομική βάση που έχουμε να έχουμε αυτούς τους δύο εταίρους, ε, συμβουλή της Ευρώπης και UNESCO. Δέκα κεφάλαια λοιπόν. Engagement, ε, δέσμευση. Πώς θα τους ε, φέρουμε πιο κοντά τους νέους, τους μαθητές, τα σχολεία, να γνωρίσουν καλύτερα την πολιτική κληρονομιά. Δεύτερο, δεύτερη δέσμη σχεδίων, βιωσιμότητα είναι ο τίτλος. Δηλαδή εδώ βλέπουμε το βιώσιμο τουρισμό, το βιώσιμο πολιτιστικό τουρισμό και πώς η πολιτική κληρονομιά μπορεί να συνεισφέρει στην αναζωογόνηση κάποιων πόλεων και περιφερειών. Όταν δηλαδή κάποια βιομηχανικά ή θρησκευτικά κτίρια μπορούν να ξαναχρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο της πολιτικής κοινωνίας. Το τρίτο είναι η προστασία. Τρίτο κεφάλαιο. Προστασία σημαίνει ε, εξορισμού, εκφύσεως, ε, πολιτική κληρονομιά. Εδώ λοιπόν έχουμε εμπλατική πρωτοβουλία για τα πρότυπα παρέμβαση ιστορικά κτίρια. Οι διεθνοί κανόνες είναι λίγο παρχιωμένη από τη δεκαετία του 1960. Πρέπει να τις φρεσκάρουμε αυτές τις, ε, αυτούς κανόνες. Και επειδή υπάρχουν πολλά ιστορικά μνημεία και κτίρια, τα οποία αναπαλαιώνονται με, με κονδύλια από τα διευθυντικά ταμεία κυρίως, θέλουμε να έχουμε ένα λόγο στο έργο που θα ξεκινήσει. Ε, πάντα στο κεφάλαιο προστασία έχουμε και κάποιες πρωτοβουλίες για να συνεχίσουμε τον αγώνα μας κατά το παράνομο, την παράνομη διακίνηση καλλιτεχνικών έργων. Και το άλλο μεγάλο κεφάλαιο είναι η καινοτομία. Τι αρμοδιότητες και ικανότητες σχετίζονται με την κληρονομία, για την διατήρηση και τη μεταφορά στις επόμενες γενιές. Κάτι πολύ σημαντικό. Και γιατί η κληρονομιά σημαίνει και οικονομικά έσοδα στην καινοτομία. Θα δούμε ό,τι έχει να κάνει με συμμετοχική διακυβέρνηση και διαχείριση, κοινωνική καινοτομία, στο πλαίσιο της σύμβασης του ΦΑΡΟ του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τέλος, η μεγάλη, ε, τελευταία μεγάλη εμβληματική πρωτοβουλία είναι να τονίσουμε την πρόοδο που έχει επιτελεστεί στον τομέα της πολιτικής κληρονομιάς χάρη στη χρηματοδότηση ε, από το ερευνητικό πρόγραμμα της ΟΠΕΞΕΜΣ. Πάρα πολύ σημαντική χρηματοδότηση. Διάφορα ε, πεδία καλύφθηκαν και δεν είναι γνωστό αυτό. Υπήρξαν μάλιστα και ανακαλύψεις που έγιναν χάρη στα ερευνητικά προγράμματα που έχουμε χρηματοδοτήσει. Και θα διοργανώσουμε ένα συνέδριο το Μάρτιο του 2018 εδώ στις Βρυξέλλες για το θέμα αυτό μαζί με τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ έρευνα. Και ολοκληρώνοντας, επανέρχομαι στην ερώτηση της κυρίας Κώστα για το πώς συνεργαζόμαστε με τις άλλες γαμαδέλτα. Συνεργαζόμαστε εντατικά. Είχαμε τρεις συναντήσεις, 13 περίπου είναι οι γαμαδέλτα που συμμετέχουν πιο ενεργά στο έργο μας για το ευρωπαϊκό έτο, έτος. Τρεις συναντήσεις λοιπόν είχαμε, πολύ θετικές, πάρα πολύ θετικές. Δεν είναι πάντα εύκολο βέβαια, όπως ξέρετε, να συνεργάζονται τα διάφορα διοικητικά τμήματα με τη ΓΔ έρευνα. Είδαμε ότι έχουμε 200 εκατομμύρια αξίας ε, ε, project που πρέπει να προωθήσουμε με τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ περιβάλλον. Είπαμε ότι θα αναφέρεται στο σχέδιο δράσης που ενέκρινε η Κομισιόν τον Απρίλιο για το Ευρωπαϊκό Έτος, για το Natura 2000. Ε, Γιατί και η φυσική κληρονομιά περιλαμβάνεται στην πολιτιστική κληρονομιά. Και με τη ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ HOME, και εδώ σταματώ, πετύχαμε το Ευρωπαϊκό Έτος να αναφερθεί στην προκήρυξη διαγωνισμού ε, στο πρόγραμμα Ευρώπη για τους πολίτες που προκήρυξα. Και είμαι έτοιμη να απαντήσω και σε οποιαδήποτε άλλη ερώτηση. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την παρουσίαση των 10 αυτών project. Πολύ καλά μου ακούγονται όλα αυτά. Για να προσπαθήσουμε να προωθήσουμε λίγο και το συντονισμό μεταξύ των κρατών μελών, αν θέλουμε να πετύχουν αυτές τις πρωτοβουλίες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ αυτή την παρουσίαση. Μου ήρθε και μια άλλη ιδέα σε ό,τι αφορά την επικοινωνία Έχουμε κι εμείς ε, το τμήμα επικοινωνία και κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε. Θα μπορούσαμε να έρθουμε σε επαφή λοιπόν μαζί σας για να δούμε πώς εμείς από την πλευρά του Κοινοβουλίου θα μπορούσαμε να προωθήσουμε και εμείς πιο εμφατικά ε, και να προβάλλουμε με τις δημοσιεύσεις μας ίσως εδώ ε, το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτικής Κληρονομιάς αν δεν έχουμε τα ευκαιρία αποτελέσματα ήδη, να έρχομαι σε επαφή. Και μια ερώτηση έχω για την άειλη κληρονομιά. Τι γίνεται με αυτό? Yeah. Non, tout à fait. Le, patrimoine η άειλη κληρονομιά είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι τμήμα των ανησυχιών μας. Θα σας δώσω κάποια παραδείγματα. Η πολιτιστική κληρονομιά που είναι άειλη είναι ακριβώς ε, η γνώση, η τεχνογνωσία και αυτό είναι και το νόημα αυτού του ε, προγράμματος για τις ε, ικανότητες, δεξιότητες. Θέλουμε και αυτή η διάσταση να εκπροσωπείται. Επίση, σε όλα τα προγράμματα που θα γίνουν ε, με τα σχολεία, με του νέου, αυτή η διάσταση τη άειλη κληρονομιά θα είναι <laughs> πολύ έντονη. Οι παραδόσει, η γαστρονομία, ο τρόπο ζωή μα, ε, ο τρόπο με τον οποίο μοιραζόμαστε ένα γεύμα, όλα αυτά είναι τμήμα τη ταυτότητά μα, τη πολιτιστική κληρονομιά μα και ενδεχομένω και των αξιών μα. Και πρόκειται λοιπόν για στοιχεία τα οποία θα ε, είναι παρόντα σε όλε τι τη συνεργασία μας με ε, στο πλαίσιο των προγραμμάτων ε, η, τα πολιτιστικά, ε, η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι και η καθημερινή ζωή, δεν είναι μόνο κάστρα που είναι απλώς κονισμένα. Γι' αυτό ακριβώς θα ασχοληθούμε και με το θέμα της άειλης κληρονομιάς. Υπάρχουν πάρα πολλά ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την άειλη κληρονομιά και με πολύ χαρά θα θέλαμε να έρθετε στη διάσκεψη που θα γίνει το Μάρτιο για το θέμα αυτό και η ταυτότητα, η οπτική ε, την οποία επεξεργαζόμαστε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους. Ε, δεν ε, μπορώ να σας την παρουσιάσω ακόμη, γιατί ακόμη την επεξεργαζόμαστε και την επαληθεύουμε. Θα δείτε όμως ότι αφορά τις εικόνες που θα χρησιμοποιηθούν και οι εικόνες αυτές θα συμπεριλαμβάνουν όλες τις πτυχές κληρονομιάς και τις άλλες. Η κυρία Κώστα. Καλλιτέχνε, μουσική, θέατρο, είναι και, και η καλλιτεχνική έκφραση, ο, ο, η, άειλη, η πολιτιστική κληρονομιά. Ναι, ναι, ευχαριστώ κυρία ε, Κώστα για την υπενθύμηση αυτή. Συμφωνούμε απολύτω και ε, θα θέλαμε να έχουμε μια σειρά προγραμμάτων ε, που μεταγράφουν τον τρόπο με τον οποίο η πολιτιστική κληρονομιά τροφοδοτεί τη δημιουργική έκφραση. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα θέλαμε βεβαίως να υποστηρίξουμε. Θερμές ευχαριστίες. Νομίζω ότι μπορούμε να σας απαλλάξουμε σήμερα. Ε, σίγουρα θα τα ξαναπούμε θα ξανασχοληθούμε με το Ευρωπαϊκό Έτος 2018 και σε όλη τη διάρκεια του έτους αυτού βέβαια που έχουμε πολλές δραστηριότητες και εμείς στις πατρίδες μας, ε, στις πόλεις μας. Μέχρι τότε βέβαια έχουμε δουλειά να κάνουμε και εμείς και εσείς. Ε, σας ευχαριστούμε και πάλι. Καλή επιτυχία και όπως είπα ε, θεωρήστε ότι στο πρόσωπό μας θα βρείτε έναν πιστό σύμμαχο πάντοτε, παρότι μπορεί να έχουμε και τη μία ή την άλλη κριτική παρατήρηση να κάνουμε. Πάντως, ο ρόλος μας ως Κοινοβουλίου και τα καθήκοντά μας τα λαμβάνουν πολύ σοβαρά υπόψη και θα, μας, ε, θα σας βοηθήσει. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι κάνετε πολύ καλή δουλειά Ελπίζω να μην το πήρατε στραβά. Απλά θα πρέπει κάποιε φορέ να ρωτάμε και εμεί τι γίνεται με τα χρήματα που έχουν διατέθει. Νομίζω είναι θεμητό από πλευρά μα Δεν έχει να κάνει με καμία διάθεση κριτική τη δουλειά που κάνετε εσεί. Απλά πάντα θέλουμε και εμείς να έχουμε ενημέρωση για το τι γίνεται με τον προπολογισμό, πώς δαπανώνται οι πόροι. Σας ευχαριστώ, καλή επιτυχία στη μελλοντική σας δουλειά και σίγουρα παραμένουμε σε επαφή. Σας ευχαριστώ που ήσασταν σήμερα εδώ.